Dear colleagues, I think we are ready to begin. Sorry for delay, but traffic in, uh, in Brussels is awful. Αυτές τις ημέρες ξέρετε ότι η κατάσταση στις Βρυξέλλες δεν είναι ομαλή. Θα περιμένουμε λοιπόν λίγο να έρθουν οι συνάδελφοι. Θα ξεκινήσω με ένα πολύ σύντομο θέμα που αφορά τους συντονιστές την χτεσινοβραδινή συνεδρίαση. Σας έχουμε στείλει όλους τις αποφάσεις των συντονιστών. Μπορείτε να τις εγκρίνετε. Τις έχετε λάβει όλοι. Χαίρομαι. Βλέπω ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι εγκρίνονται οι αποφάσεις των συντονιστών της ε, χτεσινοβραδινής συνεδρίασης. Σα ευχαριστώ. Και τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. που είναι η έκθεση πρωτοβουλίας για τις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητή είναι η κυρία Γιώτοβα, η είναι η κυρία Γιώτοβα, είναι εδώ, με στην αίθουσα. Θα γίνει η πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, για την έκθεση αυτή σήμερα το πρωί και βεβαίως έχουμε χρόνο έως τις 10 για να συζητηθεί αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Ο χρόνος πιστεύω είναι αρκετός για την παρουσίαση, την συζήτηση, καταρχήν από μέρους της εισηγήτριας και βεβαίως υπάρχουν και πολλοί άλλοι σκιώδεις. Θα δώσω το λόγο σε όλους και Έχουμε και την εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, από την Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική και τη Γεωργική Πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Βεβαίως, θα ήθελα καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι οι ερωινές περιοχές είναι περίπου το 30% της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ε, ο τομέας του τουρισμού και της γεωργίας είναι πάρα πολύ σημαντική για τις περιοχές αυτές. Υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τον πληθυσμό. Όπως ξέρετε, οι δημόσιες υπηρεσίες επίσης υπολείπονται σε πολλές από αυτές τις περιοχές. Και βεβαίως, σκοπός μας εδώ είναι να δούμε πώς η πολιτική συνοχή θα μπορέσει να βοηθήσει τις ορεινές περιοχές να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης. Θα δώσω όμως αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Γιώτοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το άρθρο 174 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο ε, το γνωρίζουμε όλοι αναφέρει τα εξής για να προωθηθεί η εναρμονισμένη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει τις δικές της πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής, της εδαφικής και της οικονομικής συνοχής στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι συνοχή σημαίνει μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερη έμφαση σε συγκεκριμένες περιοχές μεταξύ των οποίων οι περιφερειές ε, με μόνιμο μειονέκτημα, μόνιμα, ε, μειονεκτήματα γεωγραφικά ή άλλα Αυτέ οι περιοχέ, μεταξύ άλλων, είναι και οι ορεινέ. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει επικεντρωθεί επαρκώ σε αυτέ τι περιοχέ, τι ορεινέ περιοχέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει ότι εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αντιμετωπίζουν ε, έμεσα τα προβλήματα αυτών των περιοχών. Τι σκοπό έχει η έκθεσή μου να πραγματοποιηθεί ένα βήμα προς τεμπρός όσον αφορά αυτές τις περιοχές. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για αυτές τις περιοχές. Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες, αλλά έχουν και πολλές δυνατότητες. Ε, οι πλούσιοι, οι φυσικοί τους πόροι απαιτούν άριστη ευκαιρία για η ανάπτυξη. Οι φυσικοί πόροι αποτελούν κομμάτι της ευρωπαϊκής ταυτότητας στην πραγματικότητα και ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ουσιαστικά έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε το περιβάλλον αυτών των περιοχών καθώς και, τις, ε, και τους τεράστιους φυσικούς πόρους. Επίσης, ε, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις περιοχές αυτές ε, συμβάλλοντας την προστασία του περιβάλλοντος και αξιοποιώντας πολλές και διάφορες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη συνολική, ε, τις συνολικές οικονομικές δυνατότητες αυτών των περιοχών για να επιτύχουμε τον τελικό μας στόχο, δηλαδή τη συνοχή. Η έκθεσή μου αποσκοπεί να δώσει μια όθηση στη συζήτηση περί ε, εδαφικής συνοχής αλλά και να στηρίξει μια μελλοντική στρατηγική για τις ορεινές περιοχές. Ίσως να μην χρειαζόμαστε μια στρατηγική στην αρχή, αλλά μάλλον ένα θεματολόγιο όπως το αστικό θεματολόγιο. Αυτή τη στιγμή απέχουμε πολύ από την κατάρτιση μια στρατηγική ή ενός θεματολογίου, αλλά πρέπει να γίνει ένα πρώτο βήμα. Καλό θα ήταν να αξιοποιήσουμε την αναθεώρηση της ε, στρατηγικής Ευρώπη 2020 που θα γίνει σύντομα και στο μέλλον θα ε, επικαιροποιήσουμε το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και την πολιτική συνοχή. Ε, η Ευρώπη υπολείπεται των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, οπότε η πολιτική μας συνοχή θα πρέπει να, η συνοχή θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη στο μέλλον. Υπάρχουν μια σειρά προγραμμάτων, στρατηγικών και πολιτικών που εμέσως έχουν επιπτώσεις για τις ορεινές περιοχές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια προγράμματα όπως το LIFE ή το Ευρώπη 2020 ε, τα οποία είναι ιδιαίτερες σπουδαιότητες για τις ορεινές περιοχές. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Επιτρέψτε μου τώρα να σα παρουσιάσω κάποιε βασικέ αρχικέ ιδέε τη εκθεσή μου. Πρόκειται να γίνει μια συνάντηση με του συναδέλφου μου, όλου του και του συζητητέ. Του και ε, πολύ σύντομα. Επίσης είχα και την ευκαιρία να συναντηθώ με εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών, ε, ΜΚΟ, ε, εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών, να συζήτησα με πολλούς ενδιαφερομένους που εμπλέκονται στο πεδίο των ορεινών περιοχών. Με τις συζητήσεις αυτές ε, ορίζουμε το πλαίσιο για τον αρχικό μου στόχο, δηλαδή την εισαγωγή εγώ θα ήθελα μια ολοκληρωμένη εισαγωγή που θα παρουσιάζει μια επισκόψη των εργαλείων και των μέσων και των ε, νομικών πράξεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα μέσα και τις νομικές πράξεις ε, μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για τις ορεινές περιοχές. Θα πρέπει να αποτελέσουν αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη των ορεινών περιοχών σε θέματα περιβάλλοντος, ε, πράσινης ενέργειας, απασχόλησης και ευκαιριών απασχόλησης και όσον αφορά την πρόληψη της δημογραφικής κατάρρευσης αυτών των περιοχών. Εγώ πρόκειται να εστιαστώ σε όλα αυτά τα θέματα, μεν. Ωστόσο, δεν θέλω να εισβάλλω στο πεδίο αρμοδιοτήτων άλλων ε, επιτροπών. Άλλες επιτροπές μελετούν τη μακροοικονομική στρατηγική για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, για παράδειγμα. Εμένα ο σκοπός μου είναι να υπάρξει συμπληρωματικότητα μεταξύ των εργασιών των διαφόρων επιτροπών του Κοινοβουλίου, ώστε να καταφέρουμε να βρούμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για όλες αυτές τις περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Να καταρτήσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα μεταφραστεί σε ένα θεματολόγιο και ενδεχομένως ε, σε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Ορισμένες από αυτές τις περιοχές ε, δεν είναι διασυνοριακές. Είναι ορεινές περιοχές ε, εντός επικράτειας ενός μονοκράτους μέλου μέλους και εκεί έχουμε προκλήσεις τις πρέπει να αντιμετωπίσουν και υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες για αυτό το σκοπό. Να δώσω τώρα το λόγο στους Κιώδης. Ε, θυμηθείτε το χρονικό περιορισμό, όχι πάνω από 3-4 λεπτά. Παρακαλώ, κύριε Μπόκοβιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και καλημέρα σε όλους. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για τις ορεινές περιοχές ε, που ε, εκεί ισχύουν ιδιαίτερε συνθήκες και χρειάζεται ιδιαίτερη μεταχείριση ε, ω της εισηγητής για το ΕΛΚ. Θα έλεγα, όπω ακούσαμε ήδη και για την αρχική παρουσίαση της έκθεση ότι έχουμε 30% των περιοχών όπου ισχύουν δυσχερέστες συνθήκες και Διαφέρουν ε, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες εκεί και α, ισχύουν ιδιαίτερε απαιτήσει. Στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής ε, έχουμε νέες ευκαιρίες για να προωθήσουμε την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Το επίπεδο ανάπτυξης ε, διαφέρει από κράτος σε κράτος και άρα δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ομοιόμορφες λύσεις. Χρειαζόμαστε ενίσχυση της βασικής υποδομής στον τομέα του περιβάλλοντος των τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε ε, και νέες ευκαιρίες παραδείγματος χάρη ε, στο τομέα των ενεργειακών προϊόντων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πρόκειται για νέες ευκαιρίες σε σχέση με τις παραδοσιακές ενεργειακές πηγές και εδώ υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες ε, ούτως ώστε σε ορεινές περιοχές ε, σε δασικές περιοχές ε, να μπορέσουμε να να αξιοποιήσουμε το ανεκμετάλλευτο δυναμικό και να τροφοδοτήσουμε και άλλες συνοριακές περιοχές. Ε, στον τομέα της ψηφιοποίησης, εδώ υπάρχουν νέες ευκαιρίες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στην ε, διακομματική ομάδα ασχολούμαστε επισταμένα με αυτά τα ζητήματα. Ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι και λίγο κρυωμένος, γιατί ήμουνα και εγώ σε μια δασική περιοχή την περασμένη εβδομάδα και μάλλον εκεί την άρπαξα. Ε, στα πλαίσια της αλπικής μακροπεριοχής ε, έχουμε πολλά ειδικά σχόλια και θα τα καταθέσουμε στα πλαίσια των τροπολογιών. Ο κύριος Σίκοβιτς. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να προσθέσω κι εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Θέλουμε να συμμετάσχουμε στην κατάρτιση αυτής της έκθεσης γνωμοδότησης ε, η ε, στρατηγική για την περιοχή των Άλπαιων που πραγματεύεται η κυρία Μπρέσο, καθώς και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ορεινών περιοχών, είναι θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν όλους. Όχι μόνο επειδή είναι πυκνοκατοικημένες οι περιοχές, αλλά... Επίσης, διότι είναι δυνατή μια συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως και για τις παράκτιες περιοχές, έτσι και για τις ορεινές περιοχές, παρατηρούνται κοινά σημεία και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση για όλες τις ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν βασιστώ στην προσωπική μου εμπειρία, διότι ε, ήμουν για 12 χρόνια επικεφαλής της Ίστρια, Και ξέρω ότι για την ανάπτυξη της υπαίθρου τους λόφους, γιατί δεν πρόκειται για βουνά, ε, μπορέσαμε να προωθήσουμε δραστηριότητες όπως η γεωργία, ο πολιτισμός ή η βιοπικιλότητα. Επενδύσαμε στις υποδομές. Είχαμε λοιπόν μια σφαιρική προσέγγιση και αυτό εξασφάλισε και την επιτυχία του προγραμματός μας. Καταφέραμε ε, αυτήν την περιοχή να τη μετατρέψουμε στον πλέον ελκυστικό προορισμό της Κροατίας. Έρχονται από διάφορα μέρη της Ευρώπης να εγκατασταθούν πλέον σε αυτή την περιοχή της Κροατίας. Αν ακολουθήσουμε μια συστηματική προσέγγιση, μπορούμε με φύ τρόπο μια αραιοκατοικημένη εγκαταλειμμένη περιοχή να τη μετατρέψουμε σε έναν ελκυστικό πόλο για Ευρωπαίους πολίτες που ε, θα ήθελαν να κατοικούν σε ε, ορεινές περιοχές. Υπάρχουν ευφυείς λύσεις για τα προβλήματα των ορεινών περιοχών. Χρειαζόμαστε μόνο δράση, διότι υπάρχουν ήδη βέλτιστες πρακτικές, δεν χρειάζεται και να επανεφεύγουμε τον τροχό. Έχουμε εμπειρία σε αυτό το τομέα και πιστεύω ότι έτσι θα τελεσφορήσουν οι προσπάθειές μας. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω τον κύριο Πορέμπα από το ECR. Η κυρία Βάνα, ε, η επόμενη σχεδόν τη Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια για την παρουσίασή της. Και εγώ θεωρώ μια εξαιρετικά σημαντική αυτή την έκθεση για τις ορεινές περιοχές. Υπάρχει σαφώς ε, ανάγκη να δώσουμε μια νέα όθεση. Υπάρχουν βεβαίως πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και βεβαίως μέσω του Ίντερεγ. Υπάρχουν όμως και ε, συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία δεν αφορούν μόνο τις ορεινές περιοχές αλλά θα πρέπει να στηρίξουν προσπάθειες ανάπτυξης αυτής της ε, συγκεκριμένης ε, ε, περιοχής της Ορεινής. Μην ξεχνάμε όμως και το θέμα του περιβάλλοντος, γιατί ξέρετε ότι ιδιαίτερα για τις ορεινές περιοχές οι αλλαγές του κλίματος επηρεάζουν πάρα πολύ η αύξηση της θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων, Πρόκειται για περιοχές που ζουν από τον τουρισμό και οι συνέπειες της αλλαγής του κλίματος είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικές. Το ίδιο βεβαίως μπορεί να πει κανείς και για τους κατοίκους που ζουν εκεί, οι οποίοι παραδείγματο χάρη πολλές φορές πάσχουν από προβλήματα νερού, αλλά δεν είναι μόνο θέματα που μπορούν να λυθούν με συγκεκριμένες λύσεις που θα δοθούν μέσω προγραμμάτων και χρηματοδότησης. Πρόκειται για προβλήματα τα οποία απαιτούν βιώσιμες λύσεις. Και το θέμα του νερού και το θέμα της απομόνωσης και άλλων υπηρεσιών. Είναι λοιπόν κάτι που σαφώς ξεπερνάει τα όρια και τα σύνορα μιας συγκεκριμένη ορεινής περιοχής και θα πρέπει να τα δούμε πολύ πιο συνολικά. Εμείς σαν πράσινοι βεβαίως στοχεύουμε ιδιαίτερα κάποιες από τις προτάσεις το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης, της δημιουργίας ε, θέσεων απασχόλησης που θα διαρκέσουν, η βιώσιμη ανάπτυξη λύσεων για τον τουρισμό και βεβαίως θέματα χωροταξίας, περιβάλλοντος που οπωσδήποτε θέλουμε να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη. Όμως ε, κάποιες από τις προτάσεις μας ήδη έχουν ενσωματωθεί από την εισηγήτρια, ιδιαίτερα όσον αφορά τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, της κοινωνίας των πολιτών και βεβαίως έχουμε προτάσεις συγκεκριμένε πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια και βεβαίως προσβλέπουμε και σε περαιτέρω συνεργασία μαζί της. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, κυρία Αντινόλφη, είστε σκιώδης. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη, διότι συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπαν η συγκήτρια και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Δεν θέλω λοιπόν να επαναλαμβάνουμε διαρκώς τα ίδια επιχειρήματα. Τις επικρίσεις γνωρίζουμε. Και στη δική περιφέρεια έχουμε ζώνες ε, που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Ε, υπάρχει κίνδυνος αναχώρησης διαφύγης του πληθυσμού, μίσους του πληθυσμού. Πρέπει να αναφέρουμε όμως επίσης ότι και από φυσική άποψη είναι εύθραυστες αυτές οι περιοχές. Οπότε μια πτυχή που θα ήθελα να μην ξεχνάμε, ειδικότερα όταν θα γίνει η τεχνική προσαρμογή το 2016, αυτές οι περιοχές από το βορρά μέχρι το νότο πλήττονται από το γεωλογικά προβλήματα και είναι περιοχές που βρίσκονται μακριά και χρειάζονται ειδικότερα προσοχή, ειδικότερα όσον αφορά αυτό το θέμα των κατολιστήσεων. Οπότε ε, η δική μου ομάδα θα υποβάλει τροπολογίες ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε τον κατάλογο των σκηδιωδών. Ορισμένοι μάλιστα δεν είναι εδώ σήμερα. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Μπρέσο που ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια η οποία μας παρουσίασε ένα προσχέδιο σφαιρικό πλήρες ε, ε, για την εκθεσή της. Αναφέρθηκε πιστεύω στην πλειοψηφία των σημείων ε, που έχουν να κάνουν με το θέμα αυτό. Και εγώ, χωρίς να επαναλαμβάνω πράγματα που ήδη υπόθηκαν, θα ήθελα να εκφράσω μια σκέψη. Στην Ευρώπη, τα βουνά βρίσκονται κυρίως στο νότο της Υπήρου. Κατά παράδοξο τρόπο, λοιπόν, οι περιοχές όπου συναντώνται όλα οι πιθανές κλιματολογικές συνθήκες βρίσκονται στο νότο. Το καλοκαίρι μπορεί να κάνει πιο κρύο, στα μεγαλύτερα υψόμετρα ε, κρύο όπως μπορεί να κάνει και στις βόρειες χώρες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ιδιαιτερότητα η οποία συχνά παραβλέπεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Όταν ζει σε ορεινές ε, περιοχές υφίσταται δαπάνες πιο υψηλές, ε, διαρθρωτικά πιο υψηλές που δεν εξαρτώνται μόνο από τις ε, συνθήκες δημιουργίας εισοδήματος αλλά και από τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Χρειάστηκε πολύ καιρό για να αναγνωριστούν οι ιδιαιτερότητε των ορεινών περιοχών και να οριστούν συγκεκριμένε ε, ειδικέ πολιτικέ. Και εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίε ουσιαστικά ε, για την ένταξη τέτοιων πολιτικών για τις ορεινές περιοχές στα διαρθρωτικά ταμεία. Για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ουδέποτε υπήρξε κάποια συγκεκριμένη προτεραιότητα για τις ορεινές ε, περιοχές. Ακόμη και σήμερα, όπου βλέπουμε αυτό το θέμα που αναφέρει η συγκήτρια, την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές ε, για τις ορεινές περιοχές, και εδώ θα μπορούσε να υπάρξει μια πολύ σημαντική δέσμευση σε σχέση με άλλες περιοχές. Ε, να μην ξεχνάμε το γεγονός ότι πολλές από τις ε, ορεινές περιοχές αυτή τη στιγμή ε, με τουρισμό που βασίζεται στις χιονοπτώσεις θα χρειαστεί να συζητήσουν και να ξαναδούν πλήρως τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές. Ότι το έργο της εισηγήτριας είναι πολύ σημαντικό. Δεν πρόκειται για μια γενική πολιτική για τις ορεινές περιοχές. Απλά λέμε όταν ορίζονται οι προτεραιότητες να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όταν ζητάμε θυσίε από τα κράτη-μέλη πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι το κόστος των υπηρεσιών στις περιοχές αυτές ε, είναι αναγκαστικά υψηλότερο, ε, διαρθρωτικά υψηλότερο. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάσταση στις διαφορέ πολιτικές ε, εξοικονόμηση χρημάτων. Φυσικά εγώ θα ως εισηγήτρια της εκθέσης για την στρατηγική για τις περιοχές των Άλπαιων θα συντονιστώ με την εισηγήτρια ώστε να υπάρχει κάποια συνοχή παρότι βέβαια η στρατηγική για τις αλπικές περιοχές είναι πολύ ευρεία δεν περιλαμβάνει τις ε, κοιλάδες της Υπήρου που βρίσκονται τριγύρω απλά ε, για να συντονίσουμε τις διάφορε στρατηγικέ για τις ορεινές περιοχές. Ευχαριστούμε κυρία Μπρέσο, κύριο Μαρζέ, και ο εισηγητής για την έκθεση για τις ορεινές περιοχές. Θα θέλατε το λόγο, όχι. Ναι, μάλιστα. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη γιατί έφτασα ενώ είχε αρχίσει. Η συζήτηση δεν είναι εύκολη λοιπόν για μένα να πάρω το λόγο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να συγχαρώ ε, την εισηγήτρια για την ε, ποιότητα της ε, πρότασής της. Να πω ότι φυσικά και εξελίσσεται η εργασία για τις αστικές περιοχές, την αστική ατζέντα και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε τις πιο απομακρυσμένες περιφερειακές περιοχές, τις περιοχές της πέθρου και πολύ συγκεκριμένα τις ορεινές περιοχές που από το 2008, από το ξεκίνημα της κρίσης, έχουν υποστεί κέριο πλήγμα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει λοιπόν να τις ξεχνάμε από τις στρατηγικές τις οποίες επεξεργαζόμαστε. Πρόκειται για θέματα που αφορούν την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και φυσικά πολύ πιο ελκυστικές είναι οι αστικές περιοχές και οι πιο απομακρυσμένες, οι περιοχές ε, που έχουν και προβλήματα συνοχής, όπως οι ορεινές, πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, αλλά και από την αλλαγή του κλίματος. Οι ορεινές περιοχές φυσικά και έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος. Συγκεκριμένα η περιοχή των Άλπαιων που όπως ξέρετε έχουν υποστεί αυτές τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος και όσον αφορά το νερό αλλά και τους πάγους, τα χιονοδρομικά κέντρα, όπως λοιπόν ακριβώς κάνουμε και για τις νησιωτικές περιοχές, όπως κάνουμε και για τις πολύ απομακρυσμένες περιφερειακές περιοχές, όπως στοχεύουμε την αστική Ευρώπη με την αστική ατζέντα, έτσι θα πρέπει να μην ξεχάσουμε και τις ορεινές περιοχές. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τέσσερις εκπρόσωποι από την ε, DG Agri και την DG Regio. Ποιος θα ξεκινήσει? από την, ε, περιοχή, από την ε, DG Regio. Πολύ σύντομα θα κάνω κάποια σχόλια, να σας πω ότι η πολιτική συνοχής ε, με πολύ συγκεκριμένα μέτρα, όπως αναφέρατε, για τις ορεινές ε, περιοχές, παρέχει διάφορες δυνατότητες οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Έχουμε θέσει στόχους για τις ορεινές περιοχές που μπορούν και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη. Καταλαβαίνω ότι βεβαίως η έκθεσή σας ξεπερνάει την, την πολιτική συνοχής και βεβαίως περιμένουμε να λάβουμε την έκθεσή σας και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ μαζί σας. Να προσθέσω κάτι από την DG Agri. Να υπογραμμίσω, να υπογραμμίσω το γεγονός Ήθελα να τονίσω τη στρατηγική της Κομισιόν ειδικότερα για την περιοχή του Δούναβη, την αλπική περιοχή. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερως αυτή η έκθεση. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση με εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες και διάφορες γενικές διευθύνσεις για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή τη συνεργασία και προσβλέπουμε τη λεπτομερή συζήτηση. Mr. and thank you, Hakanen, uh, uh, from the presentation from DG. Ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις της DG Regio και η DG Agri. Τώρα έχετε το λόγο. Uh, thank you. It's Eva από from DG Agriculture and Rural Development from the Horizontal Rural uh, Εκτός μικροφωνίου Α, βρίσκομαστε εκ μέρους, ε, εκπροσωπούμε την ε, οριζόντια μονάδα οριζόντιας ε, πολιτικής. θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για αυτή την έκθεση και καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία να επιστήσω την προσοχή σας σε διάφορες ευκαιρίες που υπάρχουν ήδη στο πλαίσιο του Ταμείου ε, Γεωργίας και ε, Ανάπτυξης της Υπέθρου. Ήδη στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες των ορεινών περιοχών και τις προκλήσεις και ευκαιρίες που ανέφερα η συγκεντρική και σκιώδης τόσο όσον αφορά την αξιοποίηση των φυσικών πόρων τις ε, τουριστικές δυνατότητες, τις περιβαλλοντικές δυνατότητες και τις οικονομικές δυνατότητες των περιοχών αυτών ε, και προσπαθούμε να παρέχουμε και κάποιες ε, λύσεις στο πλαίσιο της ε, στρατηγικής ανάπτυξης της υπαίθρου στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Υπάρχει μια εργαλειοθήκη διαθέσιμη για την αντιμετώπιση των αναγκών των ορεινών περιοχών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Αναγνωρίζουμε τις φυσικούς περιορισμούς των ορεινών περιοχών στις ορεινές αυτές περιοχές με φυσικούς περιορισμούς υπάρχει δυνατότητα αντιστάθμισης των των εισοδημάτων και των επιπλέον δαπανών των γεωργών ώστε να τους διατηρήσουμε στην περιοχή μέσω μιας αεφόρου διαχείρισης της γης και αποφεύγοντας την εγκατάλειψη των γεών. Υπάρχουν και περιβαλλοντικά μέτρα επίσης που μπορούν να ληφθούν υπόψη στον προγραμματισμό των κρατών μελών. Το τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα εφόσον προγραμματιστούν από τα κράτη-μέλη και για τις δασικές περιοχές μπορεί να είναι ιδιαίτερα υποφελή. Έχουμε μέτρα υποδομών, προτείνουμε έκτακτη παροχή βοήθειας για επενδύσεις σε ορεινές περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς και μετά υπάρχει και μια δυνατότητα δημιουργίας θεματικών υποπρογραμμάτων στα κράτη-μέλη τα οποία μπορούν να εστιαστούν στην ανάπτυξη των ορεινών περιοχών. Αναφέρθηκαν ανησυχίες ε, όσον αφορά τον ευρυζωνικό τομέα για να προωθηθούν οι ευκαιρίες ε, εργασίας από απόσταση και αυτό αποτελεί κομμάτι της ε, στρατηγικής μας Επίσης ε, παρέχουμε βοήθεια στις νεοφύσεις επιχειρήσεις νέων ε, γεωργών. Οπότε να πιστεύω την προσέξη ότι ακόμη και στη ε, τρέχουσα πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου διάφορες ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος των ορεινών περιοχών. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much. Uh... Ευχαριστώ πολύ. Η συγγήτρια, όχι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την συμμετοχή σας και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την ε, έκθεση, τη συζήτηση που θα επακολουθήσει. Να διακόψουμε για λίγα λεπτά. Περιμένουμε τον Επίτροπο και βεβαίως την Επίτροπο, συγγνώμη. Έχουμε ένα τέταρτο στη διάθεσή μας μέχρι τις 10.

Υπότιτλοι i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 Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 Uh, Μπορούμε να συνεχίσουμε τώρα με την ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω την Κορίνα Κρέτσου, που είναι η Επίτροπος Αρμόδια για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Το Σεπτέμβριο είχε έρθει δύο φορές κιόλας, ε, ε, τελευταία φορά στην Επιτροπή μας και επανέρχεται σήμερα για να μας ενημερώσει για τις εργασίες της Γενικής Διεύθυνσης ένα χρόνο αφότου ε, ανέλαβε τα καθήκοντά της. Σωστά. Το 2015 ε, για την περιφερειακή πολιτική ήταν ένα ένας πολύ γεμάτος χρόνος, ε, διότι ολοκληρώθηκαν την άνοιξη εργασίες για την μεταρρύθμιση της περιφερειακής πολιτικής και με το 2015 είναι και τα 25 χρόνια των προγραμμάτων Interreg. Ε, το συζητήσαμε χθε σε σχέση και με την έκθεση πρωτοβουλίας για αυτά τα προγράμματα. Επίσης ε, υπήρξε μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για ειδικά μέτρα για την Ελλάδα Εξετάζουμε ήδη τα μελλοντικά βήματα για να απλουστεύσουμε την πολιτική και ενδεχομένως να μεταρρυθμίσουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προετοιμαζόμενοι και για τη νέα γενιά προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε με την Επίτροπο. Ως συνήθως ε, είναι πολύ φορτωμένο το πρόγραμμά της όμως. Μέχρι τις 11 λοιπόν έχουμε μόνο χρόνο. Θα της δώσω το λόγο. Θα ήθελα όμως να σας συγχαρώ πρώτα απ' όλα εξ ονόματο των μελών της Επιτροπής μας, διότι σήμερα είναι και εθνική αργία ε, για την Ρουμανία. Η κυρία Κρέτσου, ευχαριστώ, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ε, πάντοτε έρχομαι εδώ με μεγάλη ικανοποίηση και σας ευχαριστώ ε, για την ε, πρόσκληση. Το 2015 σε διάφορες συνεδριάσεις έχουμε ήδη ανταλλάξει απόψεις. Πολλές φορές συναντηθήκαμε και στα πλαίσια της Υπουργικής του Λουξεμβούργο. Νομίζω ότι σε αυτό το πρώτο, το πρώτο έτος διεκπαιρέωσης των νέων καθηκόντων μου έχω πολλά να αναφέρω για τα πεπραγμένα και να σας ενημερώσω για τις ε, προτεραιότητες για το 2016 αλλά και για τα επόμενα χρόνια. Όπως γνωρίζετε η περιφερειακή πολιτική είναι μεγαλύτερη ο μεγαλύτερος επενδυτικός στόχος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε ότι σε αυτήν την κοινοβουλευτική θητεία και στα πλαίσια της δικής μου εντολής ε, θα έχουμε πάρα πολλές καινοτομίες ε, διότι θέλουμε να υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις επί το που θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας ε, και αυτό θα γίνει χάρη στη δράση των κρατών μελών. Από κάτω προς τα πάνω είναι η προσέγγιση μας στην περιφερειακή πολιτική και ταυτόχρονα θα δοθεί όθηση έκτονα προς τα κάτω με μεγάλη αποφασιστικότητα και περισσότερο από ποτέ δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε όπως παλιά, δηλαδή ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποιοι είναι αυτοί που ουσιαστικά πληρώνουν, θα πρέπει να είναι αμοιβαίως επωφελής η στρατηγική για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πολιτικό όραμα της ε, στρατηγικής εξ αρχής ε, βασιζόταν σε τρεις ε, σφαιρικούς στόχους. Πρώτον, η μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να συνδράμει στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής Juncker, υποστηρίζοντας με στρατηγικό τρόπο την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας βιώσιμη ανάπτυξη. Δεύτερον, στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη, ώστε η πολιτική συνοχή σε να τελεσφορήσει προ όφελο όλων των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά εξίσου σημαντικό να εξασφαλίσει ε, τακτικό, επικοδηματικό και αποτελεσματικό διάλογο με τα μέλη της Επιτροπής Ρέτζη, γενικότερα με τις βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και καλή ε, συνεργασία. Η καλή αυτή εταιρική σχέση είναι υψής της σημασίας για μένα και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα συναντιόμαστε τακτικά. με το πέρας ε, του ε, τρέχοντος ε, θα κάνουμε μια έκθεση για τα τρέχοντα προγράμματα θα είναι όλα έτοιμα ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και στην υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης και της ψηφιακής ενίας αγοράς. Πέραν αυτό που γνωρίζετε έχουμε δύο μεγάλες κρίσεις ε, για την Ελλάδα η κρίση ρευστότητα και η άφηξη των, ε, ε, μαζική άφηξη μεταναστών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση και Φυσικά ε, το κομμάτι της περιφερειακής πολιτικής που σχετίζεται με αυτό είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικότερης στρατηγικής που πρέπει να ακολουθεί. Θα επανέλθω σε αυτό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας για τις τροπολογίες για την Ελλάδα καταφέραμε να μεταρρυθμίσουμε το CPR εγκαίρως για να βοηθήσουμε την Ελλάδα και στενά συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές ε, ούτω ώστε τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία στρατηγικών επενδύσεων να διοχετεύσουν τα κονδύλια εκεί που τα χρειαζόμαστε για την ε, μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Ε, τροποποιούμε τα προγράμματα αυτή τη στιγμή στο μέτρο που χρειάζεται ούτως ώστε τα κράτη-μέλη και οι επιμέρους περιοχές να είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε αυτήν την άνευ προηγούμενη προβλεπτή κρίση. Έστειλε επιστολή στα κράτη-μέλη εξηγώντα τι δυνατότητε που προσφέρουν τα ταμεία που διαχειριζόμαστε και του κάλεσαν να υποβάλουν ταχύτερο δυνατό τι προτάσει. Στου πέντε κράτη-μέλη έχουν ήδη απαντήσει στην επιστολή μου και άλλοι σκέφτονται ε, ακριβώ ε, ποια δέσμευση θα πρέπει να αναλάβουν στα πλαίσια των ταμείων. Ε, μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες συνέχεια, όπως είπα, και για την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, είναι μεικτή η διαχείριση που προβλέπεται στα προγράμματα και η επιτυχία των πολιτικής μας ε, είναι σε μεγάλο βαθμό συνάρτηση της ικανότητας που έχουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και αυτό ε, φαίνεται ξεκάθαρα σε δύο τομείς. Η Task Force για την καλύτερη υλοποίηση και οι προσπάθειες που κάνουμε για την απλούστευση και την ενίσχυση της διοικητικής μας ικανότητας. Η συγκρότηση της Task Force για την καλύτερη μεγαλύτερη υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής ήταν ε, από τις πρώτες πρωτοβουλίες που ανέλαβα όταν ε, ανέλαβα τα καθήκοντά μου και προσωπικά μετέβησα στα κράτη-μέλη, ούτως ώστε η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Ρέτζιο ε, να κάνει 70 περίπου συνεδριάσεις τεχνικού χαρακτήρα και για να καταλήξουμε σε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε κράτους μέλους. Τα αποτελέσματα της δουλειάς της Task Force ε, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και φυσικά θα σας παρουσιάσω συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία στην ε, συνέντευξη τύπου της ε, ΓΔ όταν παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της δράσης μας. Φυσικά ξέρετε ότι στην καρδιά αυτών των εξελίξεων βρίσκεται το ζήτημα της απλούστευσης, ε, της στόχευσης της πολιτικής μας, ε, ε, την οποία θέλουμε να βασίσουμε σε συγκεκριμένες επιδόσεις. Έχουμε έτσι την νέα πρωτοβουλία για την απλούστευση στην ειδική ομάδα εργασίας που συνεδριάζει για δεύτερη φορά σήμερα στην Επιτροπή. Αγαπητοί συνάδελφοι, υποστηρίζουμε τη δική σας δράση και η καλή μας συνεργασία ήταν αποφασιστική σημασία όχι μόνο για την βελτίωση της πολιτικής μας αλλά και για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων. Θα ήθελα και πάλι να σε ευχαριστήσω για το 2016. Θα ήθελα να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά και η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε μέσα σε ένα ειλικρινή, επικοδομητικό και αποτελεσματικό διάλογο με την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου. Φυσικά έχουμε συναντηθεί με τον κύριο Σούλτσο για να ορίσουμε το κοινό μας ε, θεματολόγιο ε, και ε, να θεσπίσουμε αυτή την τακτική ανταλλαγή απόψεων για το 2016. Αφήστε με επίσης να προσθέσω κάποιες παρατηρήσεις για τις προτεραιότητες για το 2016. Δύο είναι οι βασικές προκλήσεις που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, θα θέλαμε να πετύχουμε αποτελεσματική υλοποίηση των νέων προγραμμάτων εξασφαλίζοντας ότι τα συμπεφωνημένα το 2015 θα υλοποιηθούν το 2016, εστιάζοντας όλους ιδιαίτερως στις συγκεκριμένες επιδόσεις φυσικά. Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή, την υλοποίηση των προγραμμάτων. Επίσης, ε, μετά το 2020 και η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτά είναι δύο βασικά στήματα που μας απασχολήσουν. Το 2016 θα προσπαθήσουμε να απλουστεύσουμε περαιτέρω την περιφερειακή πολιτική Είχαμε έναν ιδιαίτερα εντατικό διάλογο ε, τον περασμένο μήνα για να πλουστεύσουμε την πολιτική και πρέπει να δούμε ποια στοιχεία της ε, πολιτικής μας είχαν ιδιαίτερη επιτυχία αναλύοντας έτσι τις ε, εναλλακτικές λύσεις για το 2016 βασιζόμενες συγκεκριμένα στοιχεία. Στις αρχές του 2016 θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα συγκεκριμένα μέτρα για να μειώσουμε το διοικητικό άχθος για τους δικαιούχου των ταμείων για να παρακολουθήσουμε αυτά που ήδη κάνουν τα κράτη-μέλη και να αναγνωρίσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και ελπίζουμε το ταχύτερο δυνατό να μπορέσουμε να υποβάλουμε τις συστάσεις για το 2016. Δεύτερον, ένα τμήμα της ε, απλούστευσης είναι και η ευελίξια ε, με την οποία θα εφαρμόζουμε τις ε, πολιτικές μας για να αντεπεξέλθουμε και σε μελλοντικές προκλήσεις όπως και οι τωρινές, όπως η προσφυγική κρίση. Ενισχύοντας τον τρίτο πυλώνα του ε, επενδυτικού σχεδίου και της οικονομικής διαχείρισης και ε, βασιζόμενοι σε συγκεκριμένες επιδόσεις ε, θα προωθήσουμε τις βασικές μας προτεραιότητες στα πλαίσια της 7ης έκθεσης για την πολιτική συνοχή που έχει προβλεφθεί για το 2015 για την οποία θα γίνει ευρεία δημόσια διαβούλευση. Αυτά τα στοιχεία ήθελα να αναφέρω σήμερα. Ευχαριστώ σας και πάλι για την υποστήριξή σας διότι θα είναι έτος μεγάλων προκλήσεων το 2016. Σας ευχαριστώ για την πραγματογνωμοσύνη σας και για την εμπειρία, την εμπειρία που έχετε και τη δέσμευση που δείχνετε ε, να μεταρρυθμίσετε την πολιτική συνοχή σε όφελος των πολιτών. Σας ευχαριστώ και προσβλέπουμε υπομονησία στη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επιτρόπε. Να δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής ε, Ρέιτζη και ξεκινώ από τους συντονιστές. Κύριε Βανίστελ Ρόι, ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ κύριε Επίτροπε και που έχουμε αυτή την ευκαιρία να δούμε τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι καλή στιγμή, πλησιάζουμε στα τέλη του έτους, είναι η τελευταία μας συνεδρίαση. Καταρχάς, ε, συμμεριζόμαστε την ισχυρή δέσμευση να ξεκινήσει αυτή η νέα περίοδος, να γίνει πραγματικότητα και να εφαρμόσουμε όλε αυτές τις ιδέες απλούστευσης. Τόσο η Επιτροπή όσο και εσείς και εμείς στην Επιτροπή μας ε, προσπάθουμε να εργαστούμε ε, με βάση αυτά. Θυμάμαι ότι είχαμε παρουσιάσει ένα προφορικό ερώτημα της Επιτροπής μας για την απλούστευση και του χρόνου θα προβάλλουμε το θέμα όλο και περισσότερο μέσω προφορικών ερωτήσεων που θα συζητηθούν στην Ολομέλεια ώστε να προχωρήσουμε με περισσότερες μάλιστα εκθέσεις υλοποίησης. Αυτή είναι η προσέγγιση που χρειαζόμαστε για να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά. Γιατί έχουμε το νομικό έργο αφενός, το οποίο λειτουργεί για 5-7 χρόνια και τι γίνεται στο μεταξύ, στο ενδιάμεσο. Η επόμενη έκθεση για το άρθρο 16 μας δίνει, θα μας δώσει μια καλή εικόνα για τα αποτελέσματα των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και την εκκίνηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για το επόμενο έτος και είναι μια καλή ευκαιρία για να εμβαθύνουμε ε, στα αποτελέσματα. Αναφέρατε την ενδιάμεση αναθεώρηση και το μέλλον. Να σας πω ποια είναι η δική μου αίσθηση. Η αίσθησή μου είναι ότι στην περίοδο 2007-2013 και στην περίοδο 2014-2020 έχουμε μάθει ότι αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο κατάρτισης των κανονισμών θα αντιμετωπίζουμε διαρκώς τα ίδια προβλήματα. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί δεν έχουν απορροφηθεί επαρκώ τα κονδύλια στην περίοδο 2014-2020 ήδη από τώρα. Είναι γιατί έχουμε ένα δύσκολο σύστημα. Υπάρχουν χίλιοι λόγοι. Κανείς δεν καταλαβαίνει γιατί χρειάζεται τόσος χρόνος. Αν δεν αλλάξουμε το σύστημά μας και δεν ε, χρησιμοποιήσουμε την έκθεση ε, της πολιτικής συνοχής 2007 αμέσως για τους ίδιους κανονισμούς, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Το 2017, συγγνώμη, το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο και το ίδιο θα γίνει και το 2020. Και είναι κρίμα. Σας ρωτώ λοιπόν, μπορείτε ε, να κάνετε κάποια πρόταση για την προετοιμασία αυτή τη νέα περίοδου. Έτσι θα μπορούσατε, αυτή θα μπορούσε να είναι και η κύρια σας συμμετοχή όταν συζητάμε το πολιτισμό σε νομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε διαρκώ τη συζήτηση για την πολιτική συνοχή, δεν μπορεί να περιμένει. Όσον αφορά λοιπόν την αναθεώρηση του μελλοντικού μας σχεδιασμού για την επόμενη προγραμματική περίοδο, ε, ε, κάτι τέτοιο θα είναι απολύτως απαραίτητο. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που ήθελα να εκφράσω σήμερα το πρωί. Μπορείτε να παρουσιάσετε αυτή τη νέο προγραμματισμό ε, ο οποίος πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στις ε, ταχύες μεταβολές του κόσμου σήμερα. Και τελευταία μου παρατηρήση ε, ζήτησα στις δικές υπηρεσίες να έρθουν να συζητήσουν στην ομάδα για το MFF και πάντα μας απαντούν το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι. Εμείς είμαστε έτοιμοι, αλλά εσείς δεν είστε δεν μπορούν να έρθουν οι δικοί σας ε, να μας πούν τίποτα ε, στην ομάδα υλοποίησης της Επιτροπής μας. Ε, αρχίζω να ανυπομονώ λίγο. Αναμένω μια απάντηση. Ευχαριστούμε. Κυρία Κρέλ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Κορίνα που σήμερα ήρθε για άλλη μια φορά εδώ στην Επιτροπή Φυσικά ένας χρόνος είναι πολύς αλλά και λίγος χρόνος. Έχω κάποιες ερωτήσεις που θέλω να κάνω όσον αφορά αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Θα ήθελα να ξέρω αν ε, ένα χρόνο μετά την αρχή αυτής της ε, θητείας όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν ήδη εγκριθεί, αν υπάρχουν δυσκολίες για κάποια συγκεκριμένα, σε κάποιες συγκεκριμένες ε, δυσκολίες που έχουν προκύψει. Επίσης, ε, αυτά που μας είπες ε, σήμερα το πρωί, αναφέρθηκες και στο θέμα της Ελλάδας και θα ήθελα να ξέρω για το 2007-2013 έχει κλείσει, έχει ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος, τα δύο δις δηλαδή είναι ήδη έτοιμα για να δοθούν, υπάρχουν όμως κάποιες ανησυχίες όσον αφορά την 31η Δεκεμβρίου. Θα τελειώσει γρήγορα το έτος και θα ήθελα να ξέρω αν όλα θα εξελιχθούν ομαλά ή όχι. Είχαμε με κάποιους άλλους ε, συναδέλφους μία συνάντηση με την Σλοβακική Προεδρία. Και αυτό που ιδιαίτερα με χαροποίησε είναι ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία για τους νέους με θέμα βεβαίως την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Ξέρω βεβαίως ότι δεν αφορά άμεσα το δική σου αρμοδιότητας, αλλά υπάρχουν πρωτοβουλίες που αφορούν την περιφερειακή συνεργασία, στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχουν και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων και κάθε τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε ένα βήμα πρόοδου. Αυτό που είπε ο κύριος Βανίστερ δηλαδή το θέμα του χρόνου καθώς και την προετοιμασία της μελλοντική διαρθρωτικής πολιτικής. Αυτό είναι κάτι που ιδιαίτερα μας απασχολεί, το θέμα του χρονοδιογράμματος. Υπάρχουν ε, διάφορες εκλογές και φυσικά θα πρέπει να υπάρξει και μια νέα επιτροπή. σίγουρα υπάρχουν πράγματα που επιταχύνουν τη διαδικασία και θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε. Χρειαζόμαστε αυτή τη φορά εκέρος να προετοιμαστούμε. Και όλοι ξέρουμε ότι οι ρυθμοί είναι τελείως διαφορετικοί από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Στην πράξη ξέρουμε ότι πρέπει να επιταχυνθεί η διαδικασία και αυτό είναι κάτι που θα το υποστηρίξουμε εμείς εδώ. Thank you, thank you, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρουερ, του ECR. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Όπως γνωρίζετε η μεταρρυθμίση και η επαναδιαπραγμάτευση του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται σε εξέλιξη και όσοι από εμάς ε, επιθυμούν να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι το 50% των Βρετανών αυτοί που θέλουν λοιπόν να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο ε, απαιτούν κάποιες αλλαγές. Αλλαγές όμως προς όφελος ολόκληρης της Ένωσης, όπως είπατε και εσείς. Αντί απλά να επιλέγουμε να μην συμμετέχουμε σε κάτι το οποίο ωφελεί όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς επισέρχεται σε όλα αυτά η περιφερειακή ανάπτυξη με το 33-35% του προπολογισμού είναι σημαντική διάσταση. Είναι μία από τις τέσσερις επικεφαλίδες στο επιστολής ε, του ε, Πρωθυπουργού βρίσκεται μπροστά την ανταγωνιστικότητα. Ε, γράφτηκε μάλιστα ένα έγγραφο από τον σύμβουλο του κυρίου Κάμερον πριν από μερικά χρόνια ε, ο, ένας τρόπος ώστε τα χρήματα της περιφερειακής αναπτύξης να γίνουν πιο αποτελεσματικά εστιαζόμενα σε δικαιούχες χώρες και περιοχές ε, ε, αξιοποιώντας τα χρήματα αυτά εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι υπάρχει ε, περιθώριο για πραγματική μεταρρύθμιση μετά το 2020. ώστε ε, να μην καταβάλουν ορισμένοι κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να τους επιστρέφονται ελάχιστα κονδύλια ε, και να του δίνονται οδηγίε για τι πρέπει να τα κάνουν έτσι ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα τα χρήματα και η τεχνογνωσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν εσεί ω επίτροπο θα εμπλακείτε σε αυτέ τι συζητήσει. Θα είστε ανοιχτοί και ευέλικτοι για μια πραγματική αλλαγή αντί για απλέ τροποποιήσεις στον κανονισμό μετά το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Γιάκοφτσιτς, ε, εκ μέρους της Άλντε. Ευχαριστώ. για την ε, παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι μεγάλη χαρά για μας και είναι και ίσως και ο καλύτερος τρόπος να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας. Θα ήθελα να κάνω ερωτήσεις για τρία διαφορετικά αλλά πολύ σημαντικά θέματα το θέμα της μετανάστευσης, ε, η κατάσταση των ε, μεταναστών, αυτό που μπορείτε ακόμα να κάνετε. Είπατε ότι πέντε κράτη-μέλη απάντησαν, ανταποκρίθηκαν. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτά. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δεσμευθείτε σε αυτό το τομέα και να παραμείνετε σε Είναι πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχετε να κάνετε για την Φύρομ, για τη Σερβία, έτσι ώστε ενώ πλήττονται από την κρίση αυτή της μετανάστευσης, να δούμε πώς μπορούν να μπουν σε μια προενταξιακή φάση. Η κρίση των μεταναστών πλήττει όλοι την Ευρώπη και όχι μόνο συγκεκριμένες χώρες. Αναρωτιέμαι επίσης τι ε, σκέψεις υπάρχουν όσον αφορά την απλοποίηση. Πώς θα προχωρήσουν οι επόμενες φάσεις της απλοποίησης. Εμείς ε, επεξεργαζόμαστε το θέμα αυτό εδώ στο Κοινοβούλιο και παρουσιάζουμε διάφορα στατιστικά στοιχεία φιλόδοξα τα οποία βεβαίως ε, όπως ξέρετε χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα από τους ε, δεξιούς και ακροαριστερούς συναδέλφους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τις ε, συγκεκριμένες περιπτώσεις φαλμάτων για συγκεκριμένα κονδύλια. Αυτό που κυρίως βαραίνει είναι η διαδικασίες, η περιπλοκότητα των διαδικασιών. Θα ήθελα επίσης να μας πείτε πώς βλέπετε και τις πιθανές συνεργασίες μεταξύ των ταμείων συνοχής και όλων των μέσων συνοχής, αλλά και των υπόλοιπων ταμείων όπως την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επίτροπο. Είναι μεγάλη χαρά για μας που βρίσκεστε σήμερα εδώ και πραγματικά θεωρούμε ότι η συνεργασία και ο διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επιτροπής Ρέτζι είναι εξαιρετικά ε, χρήσιμος. Περάσαμε μια πολύ πλούσια ε, χρονιά Προσπαθήσαμε να βρούμε απαντήσεις, να ανταποκριθούμε στην κρίση, στα προβλήματα και στις νέες εντάσεις. Να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε στην κρίση. Όπως έλεγα λοιπόν το 2015 το οποίο τελειώνει. Ήταν μια πολύ έντονη χρονιά και το σύνολο των ευρωπαϊκών πολιτικών προσπαθεί να βρει λύσεις που να ανταποκρίνονται στην κρίση. Πρόκειται για νέες δυσκολίες, νέες εντάσεις, όπως η ελληνική κρίση, αλλά και το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων. Πρέπει επίσης να πούμε ότι για θέματα πολιτικής συνοχής βρήκαμε τρόπους να ανταποκριθούμε, να αντιδράσουμε εγκαίρως και βεβαίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας συγκεκριμένα βρήκε τρόπους να απαντήσει με μέτρα συγκεκριμένα τεχνικά στην ελληνική κρίση αλλά και στα θέματα που αφορούν την μετανάστευση. Εγώ θα περιοριστώ σε δύο ή τρεις τομείς και θα σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Μίλησατε για το 2016 λέγοντας ότι θα υπάρξει μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να διαχωριστεί από το θέμα των προοπτικών, των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο μετά το 2020. Όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση, θα ήθελα να μου πείτε τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πρώτες αναλύσεις, τις οποίες σίγουρα διαθέτετε σήμερα, και εσείς προσωπικά πώς βλέπετε τη συνεργασία με την Επιτροπή Ρέζη σε αυτήν την ε, πολιτική. Τώρα, όσον αφορά τις προοπτικές για την περίοδο μετά το 2020, ήμασταν μαζί στο Λουξεμβούργο και είδαμε πως μία πιο βιώσιμη και ολοκληρωμένη απάντηση στην κρίση της μετανάστευσης. Το να συμπεριλάβουμε δηλαδή τις ευρωπαϊκές αξίες στην πολιτική μας είναι πάρα πολύ σημαντικά θέματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επεξεργαστεί ε, το θέμα με μία σειρά πρώτων ε, μέτρων Διαπιστώνουμε όμως σήμερα ότι δεν πρόκειται για συγκυριακή κρίση, χρειάζονται πολύ πιο μόνιμες λύσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ε, αυτό το φαινόμενο. Δεύτερον, σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές, ε, αν θέλετε, διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα μετά το 2008. και σε κάποιες περιοχές, αστικές περιοχές, διαπιστώνεται φαινόμενο πολύ έντονης ε, οικονομικής κρίσης, φτώχειας. Το ίδιο φαινόμενο φαίνεται και σε διάφορες άλλες απομακρυσμένες περιφερειακές ε, περιοχές της Ευρώπης. Γι' αυτό και το σύνολο των πρωτοβουλειών μας στοχεύουν στην αντιμετώπιση αυτής της φτώχειας και στις αστικές περιοχές αλλά και στις πολύ απομακρυσμένες ε, περιοχές. Κάτι που σίγουρα θα απασχολήσει και τις προοπτικές μετά το 20. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βανά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Πίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας σήμερα εδώ. Δεν είναι πρώτη φορά που είστε εδώ. Βεβαίως ε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον έτος. Θα περιοριστώ σε δύο τομείς. Δύο που δεν απασχόλησαν τους προηγούμενους ομιλητές. Θέλω να μιλήσω για τους πρόσφυγες, δεν είμαι η μόνη βεβαίως. Θα μιλήσω και για το θέμα της αλλαγής του κλίματος και της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην πρόσφατη συνάντηση των αρμόδιων υπουργών για το θέμα της πολιτικής συνοχής και στα πλαίσια της ΚΑΠ21 και των μέτρων για να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλλαγή του κλίματος. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι στόχοι και το ερώτημά μου είναι το εξής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς όλα αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν σε μία πραγματική δημιουργία θέσεων απασχόλησης και θα ήθελα να μου πείτε αν το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο συμπεριλαμβάνει κάποια μέτρα και κάποιες προτάσεις που να απευθύνονται στην αντιμετώπιση των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος. Και δεύτερον, την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο συζητήσαμε την έκθεση, μάλλον ψηφίσαμε την έκθεση για τις ε, περιοθεωριοποιημένες ε, κοινότητες και θα ήθελα να μου πείτε αν ε, έχετε συγκεκριμένα μέτρα για να υλοποιηθούν οι προτάσεις αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Κυρία Νταμάτο, ευχαριστούμε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την Επίτροπο που ήρθε εδώ για να μας ε, περιγράψει το έργο της για άλλη μια φορά. Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την μετανάστευση. Σήμερα μας είπατε πάλι ότι μέσω της πολιτικής συνοχής θα βοηθήσετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό. Εσείς επανειλημμένως έχετε υπογραμμίσει ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων 2014-2020 έχουν ήδη διατεθεί στα κράτη-μέλη χρηματοδοτήσεις αρκετά υψηλές και οι χρηματοδοτήσεις αυτές ε, αποσκοπούν στην υποστήριξη διαφόρων δράσεων υπέρ της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επενδύσεις για κοινωνικές ε, υποδομές, ε, υποδομές ε, υγειονομικές, σχολικές, στέγασης. Αλλά δεν κατάλαβα, αναφέρατε και το ενδεχόμενο αντιμετώπιση τη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε λόγω αυτή τη μετανάστευση στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακή συνεργασία και των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, η Κομισιόν έχει προβλέψει ειδικέ επιπλέον πρωτοβουλίε πέραν των όσων υπάρχουν ακόμα ε, αναφέρατε και μια επιστολή που έχει σταλεί στα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μα πείτε λοιπόν κάτι παραπάνω γι' αυτό ή πρόκειται για απλά τροποποίηση των ήδη των επιχειρησιακών προγραμμάτων που πρέπει να αξιολογούνται βήμα προ βήμα κατά περίπτωση ανάλογα με τι συγκεκριμένε ε, περιστάσει ε, που αντιμετωπίζει η εκάστοτε χώρα ή η περιφέρεια αυτά όσον αφορά τη μετανάστευση. Όσον αφορά την απλούστευση τώρα δεύτερον στην ιστοσελίδα βρίσκουμε ένα θεματολόγιο αρκετά ισχνό. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες ε, λεπτομέρειες όσον αφορά το θεματολόγιο, το χρονοδιάγραμμα, ε, τις συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, πότε θα μπορέσουμε να έχουμε μια πρώτη έκθεση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος ερωτήσεων των συντονιστών και δίνω τώρα το λόγο στην κυρία Επίτροπο για να απαντήσει ορισμένες από αυτές τις ερωτήσεις. Και ε, ελπίζω να τα καταφέρετε να απαντήσετε σε 10 λεπτά ώστε να μπορέσουμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους 8 συναδέλφους που ανέφεραν να θέλουν να υποβάλουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να επικεντρωθούμε στα θέματα που ακούμε επανελειμμένως. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη νέα περίοδο. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και συμφωνούμε όλοι να, η απλούστευση να, να συνοδεύει την υλοποίηση. Έχω υπόψη μου το ψήφισμα που υιοθέτησατε την περασμένη εβδομάδα και το άρθρο 16 που αναφέρει ο κ. Βανίστερο θα συζητηθεί μέσα Δεκεμβρίου. Αλλά να παρουσιάσω ορισμένα στοιχεία. Θα παρουσιάσω και εγώ ορισμένα στοιχεία ήδη την Πέμπτη. Συμμερίζομαι τι απόψει σα ότι χρειάζεται να δούμε τι διδάγματα έχουμε αποκομίσει, διότι χωρίς αυτά δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε, ε, ούτε να προετοιμαστούμε για το μέλλον. Η προετοιμασία για το μέλλον είναι κλειδί. Και όπως υπόθηκε πρέπει να ξεκινήσουμε τη συζήτηση όχι μόνο για την ενδιάμεση αναθεώρηση, αλλά και για την περίοδο μετά το 2020. Έχουμε ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αυτή τη στιγμή ακόμη αξιολογούμε την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Εγώ τη Δευτέρα θα πάω στην Επιτροπή ΚΟΜΠ όπου θα συζητήσουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 2014. Έχουμε λοιπόν ε, ε, αυτή την περίοδο που αξιολογούμε και φυσικά είμαστε όλοι ανυπόμονοι αλλά το 2017 θα είναι το πρώτο έτος όπου θα δούμε τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών τα αποτελέσματα των αλλαγών αυτών που έχουμε κάνει από κοινού το Κοινοβούλιο ε, και το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Ε, ε, φυσικά η χρονική στιγμή που θα εμφανιστεί ο κανονισμός θα εξαρτηθεί από την Κομισιόν ανάλογα με το πότε θα υποβάλει την πρόταση. Αλλά αφορά όμως και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας της απόφασης. Πιστεύω λοιπόν ότι η συνεργασία μεταξύ μας θα αποτελέσει παράγοντα κλειδί. Όπως αναφέραν η Κωνσταντζέ και η κυρία Κράελ, όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν υιοθετηθεί, αλλά εξακολουθούν να υφίστανται πολλά προβλήματα. Κατά την άποψή μου φυσικά η... Ε, ο ομαλότητα των δαπανών είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά και οι μεγάλες επιδόσεις, ε, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πώς η πολιτική αυτή συμβάλλει στην αλλαγή της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής τους, διότι μερικές φορές ε, κάνουμε το λάθος να συζητάμε περισσότερο για χρήματα παρά για τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής ε, στις τοπικές κοινότητες. Όσον αφορά την αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, το μελετάμε. Είναι πρόημο, ε, αλλά έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσει και θέλουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το τρέχον σύστημα. Να προσδιορίσουμε μαζί τα ερωτήματα κλειδιά, ε, τα ζητήματα κλειδιά που χρήζουν αλλαγή ε, και να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ρέτζη που μαχτεί και αυτή μαζί μας για την απλούστευση προσπαθώντας να βρούμε από κοινού ε, τι μπορούμε να κάνουμε. Αν το αποφασίσουμε μαζί μπορούμε να αλλάξουμε κάποιους κανονισμούς. Και αυτό πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Τώρα για την Ελλάδα, κάνετε μια ερώτηση για την Ελλάδα. Φυσικά, όπως είπα, είμαι ευγνώμων προς όλους σας που καταφέραμε να αυξήσουμε το ποσοστό συγχρηματοδότησης ε, στο πλαίσιο του πακέτου οικονομικής ανάκαμψης που διαθετήθηκε από την Κομισιόν. Ε, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε καθημερινά ε, με, στην Γενική Διευθυνσή Ρέντζο και έχουμε και ανθρώπους επιτόπου. Θα, πρέπει να δούμε πώς ε, θα, γίνει, θα εξελιχθούν τα πράγματα γιατί εμείς από πλευράς μας κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν για να υιοθετήσουμε κάποια έκτακτα μέτρα για την έκτακτη αυτή για τα έκτακτα αυτά προβλήματα αλλά με ανησυχούν κάποια μεγάλα έργα τα οποία έχουν μπλοκάρει εδώ και πολύ καιρό. Εμείς ε, κάναμε αυτή την ε, οικονομική ένεση στην ε, ελληνική οικονομία, οπότε δεν υπάρχει πια δικαιολογία καθυστέρησης των έργων αυτών όπως η αυτοκινητόδρομη στην Πελοπόννησο ή το μετρό της Θεσσαλονίκη. Είναι πράγματα που έχουν μείνει στάσιμα εδώ και πολλά χρόνια. Ας ελπίσουμε λοιπόν θα δούμε κάποια βελτίωση. Επίσης έγιναν εκτενείς συζητήσει. Ε, συζητάμε κάθε εβδομάδα με τους υπουργούς, ειδικότερα της Ελλάδας, γιατί όπως γνωρίζετε ε, η κατάσταση εκεί και το βλέπουμε όλοι στην τηλεόραση, η κατάσταση ειδικότερα στη Λέσβο και σε άλλα νησιά φυσικά είναι δραματική. Αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα όταν θα συζητήσουμε για τη μετανάστευση. Τώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο. Συμφωνώ μαζί σας ε, τα χρήματά μας πρέπει να γίνουν πιο αποτελεσματικά. Αυτός είναι ένας από τους τέσσερις στόχους μας. Και νομίζω πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε περισσότερο για τα αποτελέσματα που ήδη έχει αποδείξει ότι ε, φέρνει αυτή η πολιτική σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και ειδικότερα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές όπως αυτή από την οποία προέρχεστε εσείς όπου έκλεισαν τα ορυχεία, ε, και εμεί καταφέραμε να δημιουργήσουμε χιλιάδε νέε θέσει εργασία με τα ευρωπαϊκά αυτά χρήματα. Είμαι πεπισμένη λοιπόν ότι αυτή η πολιτική υποστηρίζει όλε τι περιφέρειε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζω κάποια περιφέρεια είτε στι κατοχώρε, είτε στο Ρωμανοβασίλειο, είτε στη Γαλλία, είτε στη Γερμανία, είτε στην Ανατολική Ευρώπη που να μην έχει υποφεληθεί. Ειδικότερα οι χώρε που βρίσκονται εδώ και 40 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι σήμερα Έχουμε την επέτειο, 40η επέτειο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχουμε αυτά στοιχεία για το τι έχει επιτευχθεί σε διάφορες περιφέρειες με ευρωπαϊκά χρήματα. Εγώ έκανα και συζήτηση, ε, συζητώ και με εκπροσώπους ορισμένων περιφερειών του Ηνωμένου Βασιλείου και μου λένε ότι η πολιτική αυτή υποστηρίζει έργα τα οποία δεν είναι βέβαια θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο. Είμαι έτοιμη λοιπόν να συζητήσω ανοιχτά μαζί σας όλα αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να σας ενημερώσω για παράδειγμα ότι χθε υιοθετήσαμε ένα πρόγραμμα ε, που θα αποτελέσει πολύ σημαντικό πυλώνα για να επιλώσουμε τα τραύματα που έχουμε στον Ευρωπαϊκό Χάρτη. Ε, η περιφερειακή πολιτική είναι κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης των λιγότερων αναπτυγμένων χωρών αλλά και να διαδραματίσει κάποιο ρόλο για την επανένωση της Κύπρου, για την οικονομική ανάπτυξη ορισμένων περιοχών και νομίζω ότι και αυτό το πρόγραμμα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ε, Βόρειας Ιρλανδίας και Ιρλανδίας ήταν σημαντικό για να υπάρξει κατανόηση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη που υιοθετήσαμε ε, αυτό το νέο πρόγραμμα για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθούμε να διατηρούμε τη δεσμευσή μα και θα γίνουν και κάποιε επίσημε επισκέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο του χρόνου και εγώ είμαι έτοιμη να συζητήσω για το πώ θα μπορέσουμε να να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να δούμε πώς θα συμβάλλουν τα δικά μας κονδύλια σε όλα αυτά. Όσον αφορά τη μετανάστευση, ε, είχαμε ένα ερώτημα από τον κύριο Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το ερώτημα. Είναι ένα ερώτημα που βρίσκεται στα χιλιόλων και Πρέπει να σας πω ότι από την αρχή αρχίσαμε να εξεταζούμε το πώς θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε, να συμβάλλουμε και εμείς και με τη συναδέλφα μου τη Μαριάννη Τισεν ήδη από τις πρώτες εβδομάδες του φθινοπόρου συναντηθήκαμε με κάποιες αρχές για να τους πούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να συζητήσουμε και φυσικά ένα εύλογο ερώτημα ορισμένων κρατών μελών και ορισμένων περιφερειών ήταν το εξή, αν αρχίσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα και μετά έρθουν οι ελεγκτέ, και μας πούν ότι δεν είναι επιλέξιμο αυτό που κάνουμε. Κάναμε λοιπόν κάποιες συζητήσεις με κάποιους ελεγκτές και στείλαμε μια πολύ σαφή επιστολή στα κράτη-μέλη όπου είχαμε προσδιορίσει από κοινού με τους ελεγκτές τι μπορεί να γίνει και τι είναι 100% επιλέξιμο στο πλαίσιο των κανόνων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Διότι δεν χρειάζεται αλλαγή των κανόνων. Υπήρξαν κάποιε ιδέε για κάτι τέτοιο, να δημιουργηθεί ένα άλλο θεματικό στόχο για τη μετανάστευση, αλλά κατά τη δική μου προσωπική άποψη κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο. Τα κράτη-μέλη είναι εκείνα τα οποία θα αποφασίσουν κατά πόσο θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα που του έχουν διατεθεί. Αλλά φυσικά από την αρχή ε, είχαμε θεωρήσει ότι ένα τέτοιο ταμείο μετανάστευση και ασύλου θα μπορούσε να λειτουργήσει ω ε, τα, ταμείο αντιμετώπιση κατε, ε, καταστάσεων αλλά εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και ήδη έχουμε συζητήσει. Η Ιταλία ήταν η πρώτη που ήθελε να αλλάξει το πρόγραμμα. Εμείς έχουμε αποδεσμεύσει ήδη 220, 220 εκατομμύρια για το πυλώνα μετανάστευση και το είπε και η κυρία Νταμάτο ήδη. Μπορούμε να φτιάξουμε έτσι νοσοκομεία, να υπάρχει πόσιμο νερό, αλλά κάποιες χώρες δεν επιθυμούν ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά για αυτό το σκοπό. Και εγώ έκανα συζητήσεις και με το Υπουργείο της Ελλάδα, για παράδειγμα. Είναι απαράδεκτο κατά την άποψή μου να βλέπουμε τις εικόνες που βλέπουμε στην τηλεόραση. Εγώ μίλησα με τον Επίτροπο Ανδρουκαίτης που βρέθηκε στη Λέσβο σε μία μέρα έφτασαν άνθρωποι από την Τουρκία και από τη μια μέρα στην άλλη πέθαναν ε, παιδιά λόγω υποθερμίας. Πρέπει να αναλάβουμε επίγουσα δράση, επιτόπου. Χρειαζόμαστε από κάθε χώρα κάποιο έγγραφο, μια-δυο σελίδων, κάποια επιστολή που να μας λέει τι χρειάζεται να γίνει και να αποφασίσουμε από κοινού. Ε, να δούμε τι γίνεται μέσω της Frontex, δεν μπορούμε να κάνουμε μέσω του ERDF, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Βλέπουμε ήδη ότι αυτές οι επικρίσεις, ότι στην Ιορδανία ή στην Τουρκία οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζονται καλύτερα από ότι στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ε, δεν είναι φυσιολογικό. Στη Λέσβο, για παράδειγμα, υπάρχουν δύο γιατροί μόνο στο νησί. Τα χρήματα λοιπόν δεν είναι το παν. Πρέπει να ανταλλάσσουμε και εμπειρίες Υπάρχουν χώρες που έχουν τέτοιες εμπειρίες εδώ και δεκαετίες όπως οι κατοχώρες, η Γερμανία, η Γαλλία γνωρίζουν τι, με ποιο τρόπο μπορούν να υποδεχθούν μετανάστες. Άλλες χώρες δεν το γνωρίζουν και είμαι ευγνώμων προς χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία που ήδη έστειλαν στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη αυτά. Κατά τη δική μου άποψη λοιπόν αν τα κρατημέλη μελη θελήσουν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα για αυτούς τους σκοπούς, έχουμε ακόμα τέσσερις εβδομάδες ε, ε, για τα κονδύλια της περίοδου 2007-2013. Έχω και τη Σλοβανία και την Κροατία που ανέφεραν ότι θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν κάποια από τα υπολοιπόμενα κονδύλια του, της περίοδου 2007-2013 για αυτό το σκοπό και για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Πιστεύω ότι ε, η σημαντικότερη έννοια θα είναι η κοινωνική ένταξη, αλλά όπως είπα μπορούμε να υποστηρίξουμε και κατεπήγοντα μέτρα. Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, τα οποία αυτά θα αποφασίσουν τι θα γίνει. Εμείς δεν μπορούμε να ε, παναδιανύμουμε χρήματα με την πρότασή μας. Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα, απλά πολιτικό κατά πόσο δηλαδή κάποιο κράτος μέλος επιθυμεί ή όχι να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια. Όσον αφορά το ΕΠΑ, ε, εργαζόμαστε πολύ στενά με τον ε, Επίτροπο Χάν, που είναι και αρμόδιος όπως γνωρίζετε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε και το ρόλο της μακροπεριφερειακής στρατηγικής, διότι αυτό είναι το μόνο πλαίσιο όπου κράτη-μέλη και μη κράτη-μέλη μπορούν να παραμείνουν ε, γύρω από το ίδιο τραπέζι και να συζητήσουν για αυτή την κοινή πρόκληση. Θα βρεθούμε και στην ε, Λουμπιάνα για να συζητήσουμε για τις αλπικές περιοχές ε, και σε όλες αυτές τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές συζητάμε με τα κράτη-μέλη και τα μη κράτη-μέλη και Ψάχνουμε να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και να ενισχυθεί αυτή η συνεργασία, γιατί όπως είπα πιστεύω ότι και χώρες όπως η Σερβία, η Φύρομ, άλλες ε, θα πρέπει να λάβουν κάποια βοήθεια για την αντιμετώπιση όχι μόνο για την ε, επίτευξη του κοινωνικού κεκτημένου, αλλά και για να βρουν τρόπους επίλυσης ε, τέτοιων προβλημάτων. Τώρα φυσικά όσον αφορά τι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία ε, στο πλαίσιο όλων των διαθέσιμων ταμείων. Πρέπει να δούμε πώς θα συνεργαστούμε για το επενδυτικό σχέδιο, για παράδειγμα. Έχουμε συζητήσει και αύριο θα έχω και άλλη μια συζήτηση με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν για να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε τα ταμεία μας σε περιφερειακό, τομεακό και εθνικό επίπεδο για να υποστηρίξουμε έργα ε, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πιστεύω και εναπόκειται στις διοικητικές πιθανότητες των κρατών μελών ε, για να δούμε πώς θα μπορέσουν να συνδυάσουν όλα αυτά τα ταμεία. Ε, κύριε Μαρζέ, έχετε φυσικά δίκιο, το 2015 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Αλλά υιοθέτησαμε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα είχαμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση και εγώ βασίζομαι σε μεγάλο βαθμό στην Επιτροπή Ρέτζη ώστε να προετοιμάσουμε μαζί την ε, ενδιάμεση αναθεώρηση. Όπως είπα, θα συζητήσουμε το ζήτημα αυτό ε, στις κοινέ μας εργασίες του χρόνου. Έχουμε ήδη κάνει τέτοιες συζητήσεις και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε ήδη αυτή τη συζήτηση για την ενδιάμεση αναθεώρηση του MFF. Εμείς έχουμε ξεκινήσει το μελέτη εντός των υπηρεσιών μας ε, και με το έργο της ομάδας υψηλού επίπεδου για την απλούστευση ε, μας έχουν ζητήσει τώρα μια πρόταση ε, για τις αρχές του χρόνου και επίσης συνεργαζόμαστε στενά και με την Αντιπρόεδρο Γεωργίευα ώστε να βρούμε κάποια στοιχεία όσον αφορά τις επιδόσεις του προπολογισμού. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να από κοινού να προσδιορίσουμε και να συμφωνήσουμε ε, μέσω μιας πολιτικής συμφωνίας. Ε, να προσδιορίσουμε λοιπόν κάποια στοιχεία τα, για τα, τα οποία όλοι θα συμφωνήσουμε από κοινού ότι θα πρέπει να αλλάξουν ε, στο πλαίσιο της ενδιαμέσης αναθεώρησης. Αλλά όπως είπατε και το ζήτημα τι θα γίνει μετά το 2020 είναι πολύ σημαντικό και η συζήτηση θα πρέπει να ξεκινήσει το 2017 εντός του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν. Πώς δηλαδή, τι μορφή θα λάβει αυτή η πολιτική τότε. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένη για την αναγκαιότητα της συνεργασίας μεταξύ μας για τη μεταρρύθμιση αυτής της πολιτικής διότι έχουμε ακούσει τόσες πολλές επικρίσεις. Εγώ διαφωνώ, δεν χρειάζεται απλά κάποια μικροπροσαρμογή εδώ και εκεί. Πρέπει να συνεργαστούμε και να βρούμε νέες ιδέες ε, ε, για συμμετέχοντες, ε, για χρηματοδότες, για δικαιούχους, τι λειτουργεί, να βρούμε τι δεν λειτουργεί και να καταλήξουμε σε μια πρόταση που θα λάβει πολιτική συμφωνία για την περίοδο μετά το 2020. Γιατί αν δεν συνεργαστούμε μαζί, γιατί στο πλαίσιο της πολιτικής μεταρρύθμισης φοβάμαι ότι θα προβούν σε αυτή τη μεταρρυθμίση άλλοι στη θέση μας. Όσον αφορά την εδαφική πτυχή, Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς την Λουξεμβουριανή Προεδρία που έχει συμπεριλάβει στο θεματολογιό της αυτή την εδαφική διάσταση. Διότι φυσικά ε, όλοι μας είμαστε επηρεασμένοι από την περιοχή όπου ζούμε. Δεν είναι το ίδιο να φτιάχνει κανείς μια επιχείρηση σε μια αγροτική και μια αστική περιοχή, σε μια πολυπληθή, σε μια ε, αραιοκατοικημένη περιοχή. Και φυσικά και η αστική ένδυα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ προσβλέπω στη συνεργασία με την Ολλανδική Προεδρία για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι τους απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της αστικής φτώχειας και μια συνάντηση μάλιστα πρόκειται να λάβει η χώρα ε, στο Άμστερνταμ, από τη Ρίγα στο Άμστερνταμ, ε, για το αστικό θεματολόγιο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και όπως είπα έχω παρατηρήσει ότι πολλές χώρες ήδη έχουν αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια για ζητήματα μετανάστευσης διότι τα θέματα αυτά περιλαμβάνονται στην καταπολέμηση της φτώχειας, σε αυτό το θεματικό στόχο. Στο Βερολίνο πριν μερικούς μήνες, ε, πριν από αυτή την κρίση, ε, συγκινήθηκα από ένα πρόγραμμα οργανωμένο από Γερμανίδες ε, για μη Γερμανίδες, που συνιστάται στην παροχή μαθημάτων, και νομικών συμβουλών και τα λοιπά. Πρέπει να συνεχίσουν αυτού του είδους τα έργα, πρέπει να συνεχιστεί και η ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών. Δύο, έτσι ώστε να βρούμε νέες ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα χρήματα. Τώρα, όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η αναθεώρηση και η δημόσια διαβούλευση εξακολουθούν. Εγώ είμαι σε επαφή, θα ήθελα να ζητήσω από τις ε, διαχειριστικές αρχές και εσάς να κάνετε κάποιες προτάσεις. Καθώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πρέπει να επισημάνουμε τη σπουδαιότητα των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας. Τη συζήτηση αυτή την είχαμε στο Λουξεμβούργο μαζί με τους υπουργούς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μεταξύ Βελγίου και Γαλλίας Ε, το σύνορο είναι ολοκληρωμένο οικονομικά. Για παράδειγμα, μεταξύ Γαλλίας και Βελγίου βέβαια δεν υπάρχει γλωσσικό εμπόδιο, αλλά δεν είναι δυνατή η παροχή ε, επαγγελματικής κατάρτισης λόγω διαφορετικών νομοθεσιών ε, στην κάθε χώρα. Οπότε πρέπει να δούμε πώς θα μπορούσαμε να έρουμε αυτά τα εμπόδια. Εγώ συγκινήθηκα ε, είδα ότι στα σύνορα Γερμανίας και Πολωνίας έγιναν όλες οι αλλαγές στις εθνικές νομοθεσίες ώστε ε, να πάνε ε, φοιτητές από το Σλούμπιτσε στη Φραγκφούρτη ε, κάποιοι Εργαζόμενα κινούνται καθημερινά. Αυτό εξαρτάται από τη συνεργασία περιφερειών και εθνών και κρατών μελών ώστε να αντιμετωπιστούν αυτά τα διασυνοριακά προβλήματα που είναι υπαρκτά και φυσικά έχουμε το καταπληκτικό παράδειγμα για το πώς λειτουργεί για παράδειγμα μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας έχουμε ένα παράδειγμα νοσοκομείου όπου πάνε όλοι οι Γάλλοι και όλοι οι Ισπανοί που το επιθυμούν σε αυτό το νοσοκομείο. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες. Να μπορούν να μετακινηθούν ε, οι άνθρωποι καθημερινά από μια χώρα στην άλλη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αυτό το ζήτημα. Τώρα για την δράση για το κλίμα. Έχουμε αφιερώσει πάνω από 120 εκατομμύρια δις, λέει η ομιλήτρια, για την κλιματική αλλαγή. Έχουμε ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα για την ενεργειακή απόδοση και συνεργαζόμαστε στενά με τον Αντιπρόεδρο Σεύτσοβιτς και με τον Επιτροπό Κανιέτε για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Ε, είχαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση, έχουμε αυτή τη σημαντική συνάντηση τώρα του COP21 στο Παρίσι που θα μας βοηθήσει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τα πράγματα δεν αλλάζουν. Θα θυμάστε την πρώτη ακρόαση της τότε ε, μέλους σας Επιτρόπου ε, Κρέτσου και τότε είχαμε ένα πρόβλημα χρόνου. Πολλές ερωτήσεις, ε, πολύ κατατοπιστικές οι απαντήσεις. Να συνεχίσουμε τώρα λοιπόν με πολύ σύντομες ερωτήσεις, λιγότερο από ένα λεπτό παρακαλώ και ξεκινάω με τον κύριο Βαν Μίλτεμπουργκ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ευτυχής που μιλήσατε για την αστική ατζέντα. Συνεργαζόμαστε και με το Λουξεμβούργο αλλά και με τη νέα Προεδρία γιατί θεωρούμε ότι όλες αυτές οι προθέσεις και της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, οι καλύτερες από αυτές όλες θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Όσον αφορά τις καινοτόμες πρωτοβουλίες και τη δυνατότητα χρηματοδότησης προγραμμάτων για τις ευρωπαϊκές πόλεις, θα ήθελα να ξέρω πόσο έχει προχωρήσει το εγχείρημα αυτό, πώς έχουν τα πράγματα. Ποια είναι επίσης η πολιτική ηγεσία, διεύθυνση για αυτήν την αστική ατζέντα. Ποιος παίζει αυτόν τον καθοδηγητικό ρόλο. Ποιος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγκεκριμένοι επιτροπή, και είναι δυνατόν να υπάρχουν αν θέλετε τέσσερις ή πέντε διαφορετικές ε, ε, ηγεσίε ή αρχές για αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα μέτρα που προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε εξάντε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη για να ολοκληρώσουν ε, την ε, επεξεργασία αλλά και να πληρούν τα κριτήρια γιατί ξέρετε ότι μέχρι το τέλος του 2016 αν δεν πληρούν αυτά τα κριτήρια δεν θα μπορέσει να στηριχτεί η πρότασή τους. Πώς επίσης μπορεί να βοηθήσει η Επιτροπή για αυτήν την πολύπλοκη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά την εργασία και του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής, να μας στηρίξετε, να μας βοηθήσετε. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζετε εσείς. Γιατί υπάρχουν σήμερα πολύ συγκεκριμένοι συνεργάτες της Επιτροπής οι οποίοι έχουν σαν αποστολή να σας στηρίξουν. Παρ' αυτά υπάρχουν <clears throat> περιοχές που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μπορείτε να μου πείτε λοιπόν επειδή ήσασταν στην περιφέρειά μου πολύ σύντομα τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα. Η επόμενη ερώτηση. Μιλάμε για την ε, ψηφιακή ατζέντα και θα ήθελα να μου πείτε για κάποιες νέες προκλήσεις όπως η κρίση των προσφύγων, το Brexit. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι και πρόσφυγες και επειδή διαφεύγουν τρομοκρατικές επιθέσεις ή επειδή ουσιαστικά πρόκειται για οικονομικούς μετανάστες έρχονται στην Ευρώπη. Εμείς στην δική μας πολιτική ομάδα έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν και πολλοί νέοι μουσουλμάνοι οι οποίοι ουσιαστικά ζουν στην Ευρώπη, ζουν στη Γαλλία και εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη θα πρέπει να προστατευθούν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, εδώ μιλούμε για κοινωνική συνοχή. Μας απασχολεί το θέμα της κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη και για μένα αυτό είναι το θέμα κλειδί. Είμαι πεπισμένος ότι δεν πρέπει να περιμένουμε το 2020, αλλά πάρα πολύ γρήγορα να μπει το θέμα της κοινωνικής συνοχής στην προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστώ, όπως είπατε. Το θέμα της υλοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το θέμα βεβαίως ε, της πολιτικής συνοχής μετά το 2020. Όπως ε, ο κ. Λουα θα ήθελα να ακούσω γιατί βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουαλία πολύ συγκεκριμένα θα πολεμήσει με κάθε μέσο για να μπορέσουμε και εμείς να διατηρήσουμε τα πλεονεκτήματά μας και να συνεχίσουμε να υποφελούμαστε. Η Ουαλία, όπως ξέρετε, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για το θέμα των διαρθρωτικών ταμείων αλλά και της πολιτικής συνοχής γενικότερα. Και βεβαίως ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια και για το θέμα της απλοποίησης. Κάθε φορά που επισκεφτόμαστε μια περιοχή, Ακούμε τα ίδια παράπονα, βλέπουμε τα ίδια προβλήματα. Πότε λοιπόν θα προχωρήσουμε στο θέμα της απλοποίησης. Είναι απαραίτητο και θα ήθελα να μας πείτε εσείς πώς ε, μπορούμε εμείς ε, σαν ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε κάποια παρακολούθηση των προτάσεών μας από την ομάδα υψηλού επίπεδου. Ευχαριστώ πολύ κυρία ένα λεπτό θα κάνω ερωτήσεις και σχόλια. Πρώτον, οι νέοι κανόνες συγχρηματοδότησης για την Ελλάδα. Είπατε ότι θα το συζητήσετε με τον Έλληνα Υπουργό. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο Υπουργός έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα της σωστής υλοποίησης, της ορθής υλοποίησης αυτών των προγραμμάτων. Εσείς τι εκτίμηση έχετε όσον αφορά, αν θέλετε, την συγχρηματοδότηση. Είναι καθοριστικό να επιληθούν αυτά τα προβλήματα υλοποίησης. Δεύτερον, όσον αφορά την διασυνοριακή συνεργασία και άλλοι συνάδελφοι έθιξαν το θέμα αυτό, Σήμερα βλέπουμε στις ε, μεθοριακές περιοχές υπάρχουν πολλές φορές δυσκολίες τέτοιου τύπου συνεργασίας. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει αυτά να ξεπεραστούν και να επιληθούν έτσι ώστε να προχωρήσουν τα προγράμματα αυτά. Και βεβαίως το τρίτο μου ερώτημα είναι το θέμα της νέας προγραμματικής περίοδου. Λιγότερο από ένα λεπτό, λέει και ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ για τη σημερινή αργία στη Ρουμανία και θα ήθελα να ε, υποβάλω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη απάντηση για τη μεταναστευτική κρίση και στο Συμβούλιο ε, αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται ένας μηχανισμός βάσει του οποίου θα τιμωρούνται τα κράτη-μέλη που δεν εφαρμόζουν σωστά αυτόν τον κανονισμό. Πώς όμως θα επιτευχθεί η υλοποίηση και θα συμμετάσχει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι Εμείς έχουμε αγωνιστεί για να μην επιβληθούν τέτοιες κυρώσεις στις περιοχές. Και δεύτερον, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς το μέλλον της πολιτικής συνοχής στα πλαίσια της Ευρώπης των δύο ταχυτήτων. Ευχαριστούμε. Ο κύριος τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Πολύ σύντομα να αναφερθώ και εγώ στην απλούστευση όπως και οι προλαλήσαντες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα στην Ευρώπη, ε, κυρίως στη Ρουμανία γιατί έχουμε χάσει 4 δισεκατομμύρια. Πρέπει όμως να μιλήσουμε και για την αποτελεσματικότητα. Το γνωρίζετε το θέμα καλά, Επίτροπε, και το έχουμε ξανασυζητήσει στη Ρουμανία. Υπάρχουν πολλά κέντρα που δεν μπορούν να λειτουργήσουν διότι ε, δεν καθίσταται αυτό δυνατό από την νομοθεσία. Δηλαδή δεν γίνεται να απασχοληθούν άτομα ε, λόγω της νομοθεσίας. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχει ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα υποχρεούνται τα κράτη-μέλη να τροποποιήσουν την νομοθεσία σε τέτοιες ε, περιπτώσεις και τι γίνεται όταν δεν μπορούν να απορροφηθούν τα κονδύλια λόγω νομοθετικών προβλημάτων. Ευχαριστούμε λέει Πρόεδρος. Πολλές ερωτήσεις, μεγάλη πρόκληση για την κυρία Κρέτσο για να απαντήσει παρακαλώ. Ζητώ Συγγνώμη που μακρηγόρησα στον πρώτο γύρο. Ήθελα να κάνω μια γενική επισκόπηση κυρίως για το μεταναστευτικό θα προσπαθήσω τώρα να δώσω πιο συγκεκριμένες και πιο σύντομες απαντήσεις. Για την αστιακή, το αστικό θεματολόγιο φυσικά είναι σημαντικό και για τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία και για το τρίο των Προεδριών και ε, περιμένουμε με ανυπομονησία και την Ολλανδική Προεδρία και τη συμβολή της. Νομίζω ότι η αστική ανάπτυξη θα είναι προτεραιότητα ε, για την ε, Ολλανδία. Το Μάρτιο έχουμε τη σύσκεψη των δημάρχων Το, το αστικό φόρουμ επίσης ε, Τρεις θα είναι συνολικά οι εκδηλώσεις της Ολλανδικής Προεδρίας για το αστικό θεματολόγιο. Ξέρετε πως για πρώτη φορά οι πόλεις λαμβάνουν άμεσα την επιδότηση. Είναι θέμα ε, εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της ε, πόλεις. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα. Σε σχέση τώρα με το ποιο θα είναι επικεφαλής, ο Αντιπρόεδρος ο ε, και ο κ. Σεύκοβιτς ε, έχουν τεθεί επικεφαλής. Η ΓΔΡ φυσικά συμβάλλει καθοριστικά γιατί ε, μην ξεχνάμε ότι είναι και στον τίτλο, έτσι είναι ε, γάμα δέλτα περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με τους δύο συναρμοδίους αντιπροέδρους. Ω προ την απορρόφηση των κονδυλίων. Ναι, είναι κυρίω θέμα ε, διοικητική ικανότητα ε, αυτό το διαπιστώνω στις επισκέψεις που κάνω. Ε, ορισμένες φορές αυτό ο παράγοντας είναι και πιο σημαντικός από τα διαθέσιμα κονδύλια. Αυτό το στοιχείο θα το προωθήσουμε και στα πλαίσια της μεταρρύθμισης. Ε, η εξάντε αίρεση είναι ε, ιδιαίτερα σημαντική Ε, επίσης έχουμε και μία μελέτη για τις ε, μακροπεριοχές. Ήμουν στην Καμπανία και πήγα και ε, ασχολήθηκα με τα προγράμματα για τη μείωση του χάσματος ανάμεσα στο Βόρειο και στο Νότο στην Ευρώπη αλλά και ανάμεσα στις διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Υπάρχει και το σιδηροδρομικό πρόγραμμα από την Νάπολη μέχρι τον Πάρη που θα προωθήσει την ανάπτυξη όχι μόνο από το ε, βορρά μέχρι τον νότο, αλλά και ιδιαίτερα θα προωθήσει την ανάπτυξη του νότου της Ιταλίας αλλά φυσικά πρέπει να ενισχύσουμε τη ε, το διοικητικό δυναμικό, διότι στο Νότο συνιστά μεγάλο πρόβλημα. Επίσης οι παρατυπίες ε, ως προς τις δαπάνες είναι άλλο σημαντικό πρόβλημα. Περιμένουμε τον οικονομικό έλεγχο για τα αποτελέσματά του. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα συνεργαζόμενοι πολύ στενότερα με τους οικονομικούς ελεγκτές. Ορισμένες φορές ε, μας κατηγορούν ότι είμαστε στη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο πολύ πιο επίοικη σε σχέση με το ελεγκτικό συνέδριο. Δυστυχώς στην Ιταλία και λυπάμαι που το λέω κυρίως στην Νότια Ιταλία είναι σοβαρό το πρόβλημα ε, των ελλείψεων στη διοικητική δομή και των παρατυπιών. Ο υπουργό Δεβίου και Ντεβινσέντσια έχουν κάνει πολύ σοβαρές προσπάθειες για να ε, υπερπηδήσουν αυτό το πρόβλημα που φυσικά είναι ιστορικού πλέον χαρακτήρα. Δεν άρχισε ε, τώρα τελευταία να μας απασχολεί. Κύριε Μπόκοβιτς, ε, σωστά τονίσατε πόσο προβληματικό τη είναι κατάσταση για το μεταναστευτικό, η ενσωμάτωση των ε, μεταναστών και κυρίως στην αγορά εργασίας ε, είναι στοιχείο κλειδί και σε ορισμένες περιοχές η διακριτική μεταχείριση και η αποξένωση, σε αυτών των ανθρώπων είναι το πρόβλημα, όπως και εδώ στο Βέλγιο ή σε κάποιες πόλεις της Γαλλίας, ε, σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Πολύ δύσκολα μπορούν να ενσωματωθούν μετανάστες και φυσικά η κοινωνική συνοχή έχει ιδιαίτερη σημασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει ιδιαίτερο μεγάλο ρόλο να παίξει και εγώ ασχολούμαι κυρίως με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που όπως ξέρετε έχει την ε, βασική αρμοδιότητα για την ε, ε, πολιτική συνοχή. Δεν ξέρω αν σας παραφύρω ίσως το όνομά σας, Voin, πώς λέγεστε, Συγγνώμη. Τέλος πάντων, θα ήθελα Να πω ότι και οι πρόσωποι του Βασιλείου ε, έρχονται σε επαφή μαζί μας για τη διατήρηση τη πολιτική συνοχή, διότι υπάρχουν προγράμματα που φοβούνται ότι θα σταματήσουν, δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Για την απλούστευση ε, λαμβάνω ε, καταγγελίες και διαμαρτυρίες από παντού. Όταν βλέπω τόσες ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εγκαταλείπουν την προσπάθεια γιατί είναι υπερβολικά γραφειοκρατική και παχθή στη διαδικασία και χάνουν τελικά την χρηματοδότηση με θλίβει αυτό και ε, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε με την απλούστευση. Για την Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο. Συμφωνήσαμε φυσικά ότι είναι πολιτική απόφαση για το 100% ε, συγχρηματοδότηση δεν είναι νέα αυτά τα κονδύλια. Ε, έχει θέμα ρευστότητας όμως η Ελλάδα και τη βοηθούμε με τις ε, εμπροσθοβαρείς ε, προκαταβολές χρημάτων δηλαδή. Όμως αυτό πλέον δεν είναι δικαιολογία γιατί έχουμε ήδη συγχρηματοδότηση το 5% από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και εκταμιεύσαμε ήδη ε, προκαταβολικά τα χρήματα και περιμένουμε ε, τα αποτελέσματα από αυτά τα έκτακτα μέτρα για την έκτακτη κατάσταση που αντιμετωπίζει η ε, Ελλάδα. Τώρα, για τις ερωτήσεις ε, του κυρίου Μποστινάρου και του κυρίου Μπούντα. Θα ήθελα να φυσικά και εγώ να σας ευχηθώ ε, για τη σημερινή ημέρα. Ε, τώρα, ως προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, φυσικά εγώ ξεκάθαρα είπα ότι στον τωρινό κανονισμό δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στην χρήση των κονδυλίων, την απορρόφηση των κονδυλίων και την αποδοχή των ποσοστώσεων για τους μετανάστες. Όμως πιστεύω πως ε, είναι θέμα αλληλεγγύης, ε, αλληλεγγύης που ζητείται από κάποια κράτη-μέλη που έχουν τις μεγα... τους περισσότερους οικονομικούς πόρους. Νομίζω ότι αυτό είναι στοιχείο κλειδί και για πολλές χώρες ε, στην Ανατολική Ευρώπη ε, τα τελευταία 25 χρόνια είδαμε έμπρακτες εκδηλώσεις αλληλεγγύης και ορισμένες φορές οι ανατολικοευρωπαϊκές χώρες το ξεχνούν αυτό, Ρουμανία, Βουλγαρία. Ε, για 25 ολόκληρα χρόνια ζητούσαν ελευθερία για να μπορέσουν να ζήσουν και να έχουν τις επιχειρήσεις. Το ίδιο διεκδικούν και οι μετανάστες. Προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ιδιότητες. Θα είμαστε, οφείλουμε να δείξουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη μας. Ε, επίσης, η σύνδεση ανάμεσα στα διάφορα ταμεία και την αποδοχή ε, των ε, μεταναστευτικών ποσοστάσεων είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν με τις πολιτικές μας αποφάσεις να αποδείξουμε ότι μπορούμε να δράσουμε, δεν θα πρέπει να παραμείνουμε απαθείς. Είναι κοινέ οι προκλήσεις και ε, κοινή πρέπει να είναι και η απάντηση που δίνουμε. Ξαναλέω, τεχνικός πως δεν υπάρχει σύνδεση με τον κανονισμό, όμως είναι ηθικό καθήκον των κρατών μελών να δράσουν από κοινού, διότι είναι κοινά τα προβλήματα. Ως προς την ε, νομοθεσία τώρα, για το επόμενο στάδιο θα έχουμε νέα ζητήματα για τη νέα προγραμματική περίοδο, δηλαδή 2014 έως 2020. Πέρα από το ερευνητικό κέντρο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Μπούντα, έχουμε και άλλους τομείς όπου δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, Υπέθρου και Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης. Δεν υπήρχε λοιπόν σύνδεση ανάμεσα στα δύο ταμεία. Τώρα στη νέα προγραμματική περίοδο αλλάζουν ε, οι, οι όροι. Δεν θέλουμε να, ε, θέλουμε να αποφύγουμε την ε, κατασπατάληση των πόρων. Για τα τέσσερα δις τα οποία αναφερθήκατε είναι εξαιρετικά υψηλό το ποσό στο οποίο αναφέρεστε και θα κάνουμε Πρώτα απ' όλα μία ε, αξιολόγηση της κατάστασης. Ε, θα συνεργαστώ με τους αρμοδίους υπουργούς, αλλά νομίζω ότι κατά νότα το όριο θα είναι ένα δισεκατομμύριο και όχι τέσσερα. Σας ευχαριστούμε, Επίτροπε, για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση. Έχω, θεωρώ ότι απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε του χρόνου πλέον καλή επιτυχία ε, για τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες το 2015 και καλή χρονιά. Καλές γιορτές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και επειδή βιαζόμαστε, θέλουμε να συνεχίσουμε και με τη μερίσια διάταξη. Έσβησε το μικρόφωνο της Επιτρόπου. Φανταζόμαστε ότι εύχεται καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ. I was long. No, no, no, no, it's okay. Uh, dear colleagues, we continue now. Yes, we continue now with the, uh, our next. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο σημείο της μερισίας διάταξης. Το πρωί ήταν εύκολο, είχαμε αρκετό χρόνο. Να σας παρακαλέσω να εγκαταλείψετε την αίθουσα με ησυχία χωρίς να φωνασκείτε. Λοιπόν, πρέπει να ξεκινήσουμε το εργαστήριο για τα χρηματοδοτικά μέσα στην πολιτική συνοχή. Λοιπόν, να παραλείψω τα... την εισαγωγή γιατί δεν προλαβαίνουμε. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι έχουμε τρεις προσκεκλημένους ομιλητές, τρεις ειδικού οι οποίοι θα παρουσιάσουν το θέμα αυτό. Να ζητήσω από όλους όσοι αναχωρούν, παρακαλώ να αναχωρήσουν ταχαίως και να σταματήσουν οι συζητήσεις εδώ στις αιθούσεις. Αλλιώς θα διακόψω τη συνεδρίαση. Thank Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάποιους πολύ ενδιαφέροντες προσκεκλημένους έτοιμους να παρουσιάσουν ε, ε, διάφορες πληροφορίες για τα χρηματοδοτικά μέσα. Δυστυχώς έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, λιγότερο από 10 λεπτά για τον κάθε ομιλητή. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Λάγκρη ε, Μπιαμό, ε, αναπληρωτή τμήματάρχη, κυρία συγγνώμη, Λάγκρη. Ζητά συγγνώμη η Πρόεδρος, μπερδεύτηκε λόγω του θορύβου, η κυρία Ρέιτσελ Λάγκρη, κύριος Αλεξάνδρου Ρόους και Τζορτζιονίκος. Νίκος ε, καθηγητής ε, στο Πανεπιστήμιο ε, ε, της Ουγγαρίας. Ξεκινάμε λοιπόν με την αναπληρωτή τμήματάρχη, κυρία Λάνκρη. Έχετε το λόγο. Thank you very much indeed, Chair, and thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε που διοργανώσατε αυτό το εργαστήριο και που ζητήσατε να ξεκινήσουμε με μια σύντομη εισαγωγική παρουσίαση. Θα σας μιλήσω για την εξέλιξη του νομικού πλαισίου για τα χρηματοδοτικά μέσα κάποια εισαγωγικά λόγια για τα χρηματοδοτικά μέσα στην πολιτική συνοχή. Θα γνωρίζετε πολλοί από εσάς ότι στην περίοδο 2007-2013 αυξήθηκε ιδιαίτερα η χρήση αυτών των μέσων, ειδικότερα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και σε κάποιο βαθμό στους τομείς της αστικής ανάπτυξης και της στέγασης. Όταν Μιλάμε για χρηματοδοτικά μέσα από το 7 μέχρι το 13, μιλάμε για δάνεια, αλλά και πολλές εγγύησεις για δάνεια και επενδύσεις ε, ε, μετοχικού κεφαλαίου. Και μπορείτε να δείτε την τελευταία μας έκθεση που έχει σταλεί και που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο, την τελευταία έκθεση βάσει των ετήσιας έκθεση του 2014. Έχουμε τεράστιο αριθμό σύμβολων ε, 11 ε, εκατομμύρια για το ERDF και το DSF δεν αποτελούν αυτό σκοπό. Είναι ένας τρόπος ε, παροχής διαρθρωτικών, κονδυλίων διαρθρωτικών ταμείων. Και είχαμε και κάποια σχόλια από τους τελικούς δικαιοχούς, ειδικότερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες λένε ότι προτιμούν ένα δάνειο παρά μία χορηγία. Διότι αυτό σημαίνει ότι δεν ε, κάνουν επενδύσεις χωρίς να ξέρουν αν είναι βιώσιμες. Και φυσικά όλα αυτά χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των στόχων της πολιτικής συνοχής. Πώς θα παρέχουμε αυτά τα κονδύλια μέσω των εμπορικών ε, ε, διαμεσολαβητών όπως οι τράπεζες. Αυτό προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα και στις σημερινές συνθήκες ε, μεγιστοποιεί και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παροχή των κονδυλίων αυτών. Η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για, ως χρηματοδοτικών μέσων βοηθά στην άρση των εμποδίων ε, για τις επενδύσεις. Να σας δώσω μερικά πρακτικά παραδείγματα. Ορισμένα κράτη-μέλη, ορισμένες περιφέρειες στην Ευρώπη ε, έχουν πολύ ψηλά επιτόκια τον τελευταίο καιρό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οπότε τα διορθωτικά ταμεία βοηθούν στη μείωσή τους. Οπότε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έπαιρναν δάνεια λόγω των υψηλών επιτοκίων μπορούν τώρα να πάρουν. Ένα άλλο παράδειγμα είναι κράτη-μέλη όπου είναι υπερβολικά υψηλέ οι Δεν θέλει να διακινδυνεύσει μια τράπεζα και εκεί ε, η χρηματοδοτική αρρωγή βοηθά να μειωθούν οι απαιτήσει των τραπεζών. Αλλά υπάρχουν και κάποιε δυσκολίε ε, στην προσέγγιση αυτή να επισημανώ μία από αυτές εξισορρόπηση των στόχων δημόσιας πολιτικής με τα οικονομικά θέματα ο, λόγω του κερδοσκοπικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων των δημοσιολαβητών. Οπότε χρειάζεται περισσότερη κατανόηση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ώστε να επιτευχθεί μια καλή ισορροπία μεταξύ των δύο στόχων. Στην περίοδο 2007-2013 ε, ε, παρατηρήσαμε κάποιους περιορισμούς ειδικότερα στην πλευρά του δημοσίου που επηρέασαν την παροχή των κονδυλίων αυτή έχουν προσδιοριστεί σε διάφορες εκθέσεις του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Κοινοβουλίου. Πρώτο οι διαχειριστικές αρχές είχαν να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο μέσο παράδοσης, παροχής. Είχε χρησιμοποιηθεί σε ένα δυο κράτη-μέλη, αλλά όχι σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένες φορές λοιπόν δεν καταφέραν να το διαχειριστούν η Επιτροπή εκείνη την εποχή προσέφερε κάποιες ε, ε, κοινέ πρωτοβουλίε βοήθεια μαζί με την Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα ώστε να αντιμετωπιστούν κάποια από τα προβλήματα. Αλλά η κατάσταση διορθώθηκε μόνο μερικώ. Από πλευρά του, ε, τα οικονομικά ιδρύματα που συμμετείχαν δεν είχαν ιδιαίτερη εμπειρία στη συνεργασία με το δημόσιο τομέα. Οπότε δεν ήταν επαρκώ εξοπλισμένα για να κατανοήσουν την πολιτική και του στόχου αυτή εξ αρχή. Ένα άλλο πρόβλημα, όπως τα γνωρίζετε όσοι έχετε συμμετάξει σε αυτό εδώ και χρόνια. Ε, στην αρχή το πλαίσιο ήταν ανεπαρκές. Έλειπαν απλά στοιχεία στην αρχή. Είχαμε ελάχιστα κείμενα για τα χρηματοδοτικά μέσα στον αρχικό κανονισμό. Έλειπαν διάφορες έννοιες ε, ουσιώδους σημασία στην αξιολόγηση του κενού, ε, διάφορες, ε, διάφοροι όροι χρειάστηκε να καθοριστούν αργότερα. Άλλες έννοιες, παρακολούθηση, υποβολή εκθέσεων ε, ήταν καταλληλότερες για χορηγίες παρά για χρηματοδοτικά μέσα και θυμάμαι ότι έγιναν κάποιες προτάσεις τροποποίησης του κανονισμού και ακολούθησαν μια σειρά κατευθυντήριων εγγράφων που βοήθησαν να διορθωθεί η κατάσταση μερικώς, αλλά και με κάποιες παρενέργειε, ανεπιθύμητες ενέργειες, ότι οι διαχειριστικέ αρχέ ουσιαστικά δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σε ένα σταθερό πλαίσιο. Αυτή η κατάσταση μαζί με την οικονομική κρίση που ήρθε στην αρχή της προγραμματικής ε, προόδου είχε ω αποτέλεσμα ότι οι αποδόσει δεν ήταν πάντα αυτέ που έπρεπε να είναι. Κάποιες φορές ε, δεν έφταναν τα χρήματα ε, στο δικαιούχο τόσο γρήγορα και μερικές φορές και η πλήρης η υποβολή ολοκληρωμένων εκθέσεων δεν ήταν δυνατή. Όταν χρειάστηκε λοιπόν να προετοιμάσουμε την περίοδο 2014-2020, θέλησαμε τα διδάγματα της προηγούμενης περίοδου να ληφθούν υπόψη. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν και το έργο των συνομοθετών βασίστηκε σε αυτές τις σκέψεις να πω ότι είμαστε όλοι ευγνώμονε και στο έργο αυτή εδώ τη Επιτροπή. Κάποιο μου είπε πρόσφατα ότι για τον τίτλο 4 Είχαμε περισσότερου τριμερεί διαλόγου από ό,τι ολόκληρο το MFF. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι απλά φήμη. Ε, λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ένα από τα προβλήματα είναι, όπω είπα, δεν είχαμε ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο από την αρχή. Αυτό προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε όχι απλά περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που, την που έλειπαν την προηγούμενη φορά, αλλά αφορά και όλα τα ταμεία. Οι αλλαγέ όμω δεν είναι πάντα απλέ στην υλοποίηση. Θα μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει τι αρχέ τη προηγούμενη περίοδου φυσικά, όπω υπήρχαν στην νομοθεσία. Ε, τι κωδικοποιήσαμε εντό του κανονισμού. Προσπαθήσαμε δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ε, σταθερό πλαίσιο χωρί να δημιουργούμε νέου κανόνε. ώστε να είναι σαφής από την αρχή. Κάποια από τα στοιχεία τα οποία ανέφερα όσον αφορά τα προβλήματα, ε, έλλειψη αξιολόγησης κενών ε, δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Βοηθά στη λήψη καλών ε, αποφάσεων. Δεύτερον, η αδυναμία να φτάσουν κάποια χρήματα στις μικρομεσαίες αρχές λόγω κάποιων διαδικασιών ε, έχει βελτιωθεί και μετά τα στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων ήταν σαφή από την αρχή. Οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία και διάφορες επιλογές για την υλοποίηση των μέσων. Ε, ίσως και οι διαχειριστικές αρχές καλό θα ήταν να μπορούν να υλοποιούν, να ε, πραγματοποιούν τα δάνεια μόνες τους ε, και βάσει διαφορών πρωτοβουλειών και εισήγαμε, έχουμε εισάγει και κάποια στοιχεία που αφορούν τις πρακτικές στην αγορά επειδή αυτά τα μέσα συνήθως έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το MFF, από το ΕΤΕΤΕΣ πρόγραμμα έτσι λοιπόν χρειαζόμαστε κάποιες διατάξεις ώστε αυτά τα μέσα να μπορούν να συνεχιστούν εντός φυσικά ευλογών περιορισμών και τέλος το ζήτημα της διοικητικής ικανότητας που επαναλήφθηκε σε όλους τους τριμερείς διαλόγους και όλες τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό το σκοπό έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε κάποιες δυνατότητες ε, μέσων ε, πιο εύκολων στην εφαρμογή για τις διαχειριστικές αρχές όταν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες ικανότητες ή εμπειρία. Έχουμε ένα κόμβο γνώσης που ονομαστε FICOMPAS. Δεν, δεν σας παρουσιάσω τώρα όλα τα έργα, αλλά καλό είναι να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται διάφορα σεμινάρια ε, στα κράτη-μέλη. Ε, στο πλαίσιο του ΦΙΚΟΜΠΑΣ ε, παρέχουμε εκπαίδευση και μια ευκαιρία να απαντηθούν ερωτήσεις και να αντιμετωπιστούν κάποια από τα ερωτήματα που τίθενται. Και παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις από τις διαχειριστικές αρχές, με επίσημους και ανεπίσημους τρόπους, εκδίδουμε διάφορα κατευθυντικά σημειώματα για να απαντήσουμε τα ερωτήματα αυτά. Συμπερασματικά λοιπόν, Ευχαριστούμε ότι ε, ελπίζουμε ότι αυτή τη στιγμή το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα βελτιώσει τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων. Υπολογίζουμε να μας βοηθήσουν για αυτό το σκοπό όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι επανήλθε η πειθαρχία. Τηρήσατε πλήρως το χρόνο σας. Αυτή ήταν η παρουσίαση της Γενικής ε, Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής ε, Πολιτικής. Ο κύριος Δρόους τώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω σε αυτήν την Επιτροπή. Είμαι νομικός και είμαι ειδικό για θέματα χρηματοδότησης και Ίσως ε, δεν έχω την ε, ίδια άποψη με άλλους συναδέλφους που δίνουν νομικές συμβουλές και στηρίζουν παρόμοια χρηματοδοτικά ε, προγράμματα και μέσα. Αυτό που θα ήθελα καταρχήν να παρουσιάσω είναι ποιες είναι οι ειδικέ αρμοδιότητες, εμπειρογνωμοσύνη και ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους εμείς δραστηριοποιούμαστε. Θα αναφερθώ, αν θέλετε, σε κάποιες περιοχές όπως τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία προτίθεται να χρησιμοποιήσει περίπου το 1 τρίτο των μέσων που θα μπορούσε και ίσως αυτό θα σας ξαφνιάσει, αλλά ανησυχούν ιδιαίτερα όσον αφορά και το Horizon 2020 αλλά και το COSME προβλέπουν μια χρηματοδότηση η οποία από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσει να ε, φτάσει μέχρι αυτήν την περιοχή. Εγώ θα ήθελα εδώ πολύ συγκεκριμένα να σας πω ότι έχουμε ε, πραγματογνωμοσύνη εμπειρία για το πώς να προετοιμάσουμε αυτές τις πληροφορίες και να φτάσουν οι πληροφορίες σε αυτούς οι οποίοι τις χρειάζονται. Υπάρχει βεβαίως εδώ συμφωνία όσον αφορά το μεγάλο όφελος που παρέχουν αυτά τα μέσα για τις περιοχές στις οποίες χρηματοδοτούν. Όπως είπε και η Ρέιτσελ, η ανάπτυξη του νομικού πλαισίου είναι πολύ ορθό το ότι πραγματικά η Επιτροπή τα έχει επεξεργαστεί. Από μέρους τώρα των ε, κρατών μελών για να υπάρχουν πιο ε, γρήγορες λύσεις και καλύτερη, αν θέλετε, συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες συγκεκριμένες ε, δράσεις. Τώρα, τι πάει καλά και τι πάει λιγότερο καλά, αν θέλετε. Σίγουρα κάποιες συγκεκριμένες και σαφείς ε, νομοθετικές διατάξεις θα μπορέσουν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να έχουν πρόσβαση και να δια να περάσουν στις ε, ευρωπαϊκές αρχές τις πραγματικές τους ανάγκες. Έχουμε εδώ κάποιες ε, συγκεκριμένες, αν θέλετε, διαδικασίες τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά αυτό που σίγουρα δεν είναι βοηθητικό και χρήσιμο είναι οι πολύ συγκεκριμένες ε, νομοθεσίες, οι οποίες είναι περιοριστικές, περιορίζουν την καινοτομία, διότι βλέπουμε ότι σε αυτή την περίπτωση είναι περίπλοκα τα συστήματα και δεν μπορούν οι εταιρείε, οι φορείς του ιδιωτικού τομέα να συμπεριληφθούν σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι παράλληλα με τα μεγάλα δημόσια προγράμματα να διευκολυνθεί η συνεργασία με τις άλλες αρχές των κρατών μελών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαρθρωτικά ταμεία. Εδώ θα πρέπει να εντοπιστούν τα σφάλματα, να διορθωθούν, παραδείγματος για την περίοδο 2007-2013, η ε, λίστα, ο κατάλογος των σφαλμάτων δεν έχουν ακόμα δημοσιευθεί. Αποσαφήνιση των κανονισμών. Βεβαίω καταλαβαίνουμε ότι οι προσπάθειες της Επιτροπής να αποσαφινιστούν κάποια τμήματα των νομικών θωμάτων είναι επίσης κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί, να υποστηριχθεί. Τους ευχαριστούμε για αυτό. Αυτό όμως θα πρέπει πραγματικά να φέρει κάποια αποτελέσματα. Το θέμα τώρα της πρόσβασης στις υπηρεσίες. Δεν λειτουργεί το σύστημα top-down, από πάνω προς τα κάτω, η διάχυση δηλαδή των πληροφοριών. Και αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο, 2014-2020, σίγουρα έχουν ξεκινήσει με πολύ θετικά βήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, κρατικές επιχορηγήσεις και τις εξαιρέσεις από αυτές. Ξέρουμε ότι περάσαμε από 2,5 σε 15 εκατομμύρια για αυτήν την ε, προγραμματική περίοδο. Το άρθρο 21.13c που προβλέπει τις ε, διατάξεις για την συγχρηματοδότηση, την συμμετοχή, αυτό το 25% το οποίο τελικά δεν είναι δεσμευτικό και θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Η αρχική πόροι που θα πρέπει να διατίθεται και σε κάθε περίπτωση το κατά πόσον πρέπει η χρηματοδότηση από μέρους των κρατών μελών να γίνεται από την αρχή. Όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτά τα νέα προγράμματα 2014-2020, οι κανόνες, επαναλαμβάνω, είναι περίπλοκοι, διαρκώς αλλάζουν, ιδιαίτερα για τα διαρθρωτικά ταμεία βλέπουμε πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες και πραγματικά πολλές φορές αυτές οι τόσο περίπλοκες διαδικασίες και αυτό είναι κρίμα αποτελούν πραγματικό εμπόδιο στην συμμετοχή αυτών οι οποίοι θα ήθελαν να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση αυτή. Χρειάζονται λοιπόν σε κάποιους τομείς νέοι κανόνες, οι οποίοι όμως θα γίνουν πιο σταθεροί. Η κάθε αλλαγή που γίνεται έτσι κι αλλιώ ελέγχεται, χρειάζεται λογιστικό έλεγχο, κάτι που για μας αποτελεί μια επιπλέον διαδικασία, ένα επιπλέον γραφειοκρατικό άχθος. Αυτή λοιπόν η περίπλοκη διαδικασία, το υψηλό κόστος, σίγουρα απαιτεί περισσότερη απλοποίηση. Ολοκληρώνω. Στηρίζουμε και χαιρετίζουμε τις περισσότερες από αυτές τις αλλαγές. Βεβαίως εδώ εμείς θα προτείναμε μία περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών. Η DG Competition η οποία έχει ξεκινήσει με τη διαδικασία εξυγχρονισμού, απλοποίησης και έχουν ξεκινήσει την επεξεργασία αυτών των διαδικασιών με σκοπό να τις απλοποιήσουν και να μπορέσουν να καλύψουν περισσότερα προβλήματα. Το κάθε κράτος μέλος βεβαίως έχει ένα σημείο επαφής για την πρόσβαση σε αυτές τις διαδικασίες. Εμείς ε, θα θέλαμε αυτό να διευρυνθεί και να επεκταθεί στο μέλλον. σε ευχαριστούμε και τώρα πάμε στον επόμενο μιλητή, την κυρία Νίκολς από το ε, Εθνικό Πανεπιστήμιο Δημοσίων Υπηρεσιών της Ουγγαρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω την η ε, ικανοποίησή μου για τη σημερινή πρόσκληση για να σχολιάσω ε, κάποια ε, χρηματοδοτικά μέσα, κυρίως το τη συνδυασμένη μικροπίστωση, ένας μηχανισμός που υπάρχει στην Ουγγαρία δηλαδή, για την δημιουργία, ε, την επιβίωση και την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, ένα στοιχείο κλειδί ήταν η μικροπίστωση. Είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο. Πρόκειται για αρρωγή ε, που μπορεί να ζητήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν επιστρέφεται η επένδυση. Χρησιμοποιείται λοιπόν αυτός ο μηχανισμός στην Ουγγαρία. και ε, είμαστε και πρωτοπόροι στην Ευρώπη. Όπως ακούσαμε, ε, τα χρηματοδοτικά μέσα λόγω του στοιχείου του revolving ε, της επιστροφής επένδυσης δηλαδή έχουν ιδιαίτερη σημασία με την οικονομική κρίση και σήμερα τα χρηματοδοτικά μέσα είναι ένας τομέας ε, που ε, ελκύει το ενδιαφέρον αυτών που καταρτίζουν την πολιτική και σε κυβερνητικό επίπεδο. Το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ευρώπης αναφέρει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την υλοποίηση σταδιακών επενδύσεων. Η πρακτική στην Ουγγαρία, λοιπόν, το 2004 στο 2006 Τα προγράμματα έτρεχαν χωρίς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, όμως για την περίοδο μέχρι το 2013 άλλαξε η κατάσταση. Για την περίοδο 2007 2013 ε, όταν βλέπουμε τα ποσά ε, ως ποσοστό του, της περικοδότησης ε, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ανερχόταν στο 6% και για τα επιχειρησιακά προγράμματα αυξήθηκε κατά 30% η στήριξη μέσω τροποποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπου Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και η Ουγγαρία αποφάσισε το 2007 να υλοποιήσει το Τζέρεμι χωρίς ε, ε, ενωσιακή χρηματοδότηση, χρησιμοποιώντας μόνο ε, PRC επιχειρηματικού κεφαλαίου. Τα χρηματοδοτικά μέσα μπορούν να είναι πολύ περίπλοκα ε, και χρειαζόμαστε γι' αυτό διαχειριστικές ομάδες εμπειρογνωμόνων. Ε, χρησιμοποιούμε το ε, λυσιδωτό σύστημα, δηλαδή επιλέγεται από το διαχειριστική αρχή ο διαχειριστής του holding fund και στη συνέχεια γίνεται υποβολή πρόσκλησης προσφορών για τους διαμεσολαβητές. Προτού φτάσουμε στους δικαιούχους επιτόπου μέσω των χρηματοδοτικών μέσων. Θα πρέπει όμως να αναφερθώ και σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε κατά την προετοιμασία του συστήματος των ε, χρηματοδοτικών μέσων αναρωτηθήκαμε αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ε, κρατικές προμήθειες για την επιλογή των διαμεσολαβητών ή όχι. Βάσει του κανονισμού για την πολιτική συνοχή ε, θα πρέπει να επικρατεί διαφάνεια και να είναι ανολογικά οι διαδικασίες ώστε να αποφεύγονται ε, οι συγκρούσει συμφερόντων, αποκλείοντας έτσι de facto τις κρατικές προμήθειες στην Ουγγαρία για την περίοδο 2007 έως 2013 έτσι είχε η κατάσταση, όμως ε, πρόσφατα μάθαμε το αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους κανόνες για τις κρατικές προμήθειες. Είναι διαφορετική η ερμηνεία του κανονισμού, δηλαδή στην περίοδο 2007 έως 2013 η διατύπωση δεν έχει αλλάξει και σας διαβεβαιώ πως το ουγγρικό σύστημα εξασφαλίζει ε, μία λύση. Ε, μετά από το holding fund έχουμε ολόκληρο δίκτυο με σε οικονομικούς διαμεσολαβητές και βάσει του κανονισμού αυτοί οι διαμεσολαβητές πρέπει να προσθέσουν ε, στο ταμείο τα δικά τους κεφάλαια σε περίπτωση ε, χρηματοοικονομικών ε, οργανισμών το ποσοστό είναι τουλάχιστον 25%. Σε περίπτωση οργανισμών μικροπίστης ε, είναι το ελάχιστο ποσοστό 10%. Οι διαμεσολαβητές λειτουργούν βάσει του κέρδους ανάμεσα στη πηγή κεφαλαίων χαμηλού ε, κόστους ε, με ποσοστό 0,4% και τη διαφορά λοιπόν με το επιτόκιο που πληρώνει ο πελάτης. Δεν ε, καταγράφουμε όμως το διαχειριστικό κόστος διότι δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Για το προϊόν, να το ονομάσω έτσι, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια πώς χρησιμοποιήθηκε στην πράξη η μικροπίστη ήταν ε, για μας ένα πολύ σημαντικό μέσο. Άλλαξαν όμως τρεις φορές οι αρχικές παράμετροι του συστήματος για να ανταποκριθούμε και στην κρίση. Μετά ε, την κρίση ήταν σχεδόν αδύνατο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, να λάβουν από εμπορικές τράπεζες δάνεια. Ως πιθανή λύση σκεφτήκαμε το 2011 τα ήδη υφιστάμενα προγράμματα μικροπίστης ε, ε, συνδυάζοντάς τα με το σύστημα ε, επιδοτήσεων. Κατανότα το όριο είναι το 45% για τα δάνεια μέχρι 10 εκατομμύρια και 60% μέχρι 20 εκατομμύρια τα υπόλοιπα είναι ήδη οι πόροι, το όριο 10% της συνολικής επένδυσης. Αυτό το μίξ ε, προτείναμε. Ε, δεν μπορούμε να υπερβούμε το ποσό αυτού του κεφαλού που πρέπει να επιστραφεί και, δεν μπορούμε να, ε, και τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να είναι κάτω από το 10%. το δάνειο είναι υποχρεωτικό κομμάτι του προγράμματος το, η, η, μικροπίστη συνδυάζεται λοιπόν με επιστρεφόμενα και μη επιστρεφόμενα κεφάλαια, εξού και η, η καινοτομία αυτού του νέου συστήματος της μικροπίστης. Το μέσο επιτόκιο ε, ήταν ε, περίπου 7% για το σύνολο του προγράμματος. για εργαλεία πληροφορικής, για βασική υποδομή, κυρίως για επιχειρήσεις startup. Αυτή ήταν η στόχη μας. Έχουμε διάφορα ε, χρηματοδοτικά μέσα και κυρίως χρησιμοποιούμε συνδυασμούς αυτών ανάλογα με ε, τον οικονομικό σχεδιασμό των μικροεπιχειρήσεων. Πάντως με υποχρεωτική χρήση και χρηματοδοτικών μέσων ε, πέρα από τις επιδοτήσεις. Ε, έχουμε και ένα σύστημα μονοαπευθυντικής θηρίδας, One Stop Shop, για να βοηθούμε τις μικροεπιχειρήσεις. Μετά την τροπή των προγράμματων και την υλοποίησή του το 2007 για τα επιχειρησιακά προγράμματα είδαμε τη μεγαλύτερη πρόοδο στην υλοποίηση από πλευράς ακριβώ των μικροεπιχειρήσεων και μεγαλύτερη συμβολή σε σχέση με βασικούς δείκτες που χρησιμοποιούμε για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Η χρήση τα τελευταία τρία χρόνια ήταν 100%, ε, η απορρόφηση δηλαδή των κονδυλίων. Ε, στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές ε, είχε ειδικό βάρος αυτό το σύστημα της μικροπίστης και φαίνεται ότι στην πράξη λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ιδού τα αποτελέσματα της χρήσης των διαφόρων μέσων βασιζόμαστε σε χαρακτηριστικά όπως η στενή σχέση με τους πελάτες, η γεωγραφική κατανομή και η στο ότι ε, η χρηματοδότηση συνδυάζεται με επιδοτήσεις που λαμβάνουν σε άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το βλέπετε αυτό στη διαφάνεια. Το μεικτό αυτό σύστημα είναι πάρα πολύ ευνοϊκό για τις ε, περιοχές στην Ήπεθρο, για τις γυναίκες ε, και βλέπουμε ότι ακόμη και σε προβληματικές λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές έχει ε, ιδιαίτερα ωφέλη. Ε, κίνδυνος οικονομικού ελέγχου τώρα που συνδυάζεται με το μεικτό σύστημα μικροπίστης. Όπως σας είπα, συζητήσαμε ε, ε, εκτενώς με τις ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να συμμορφωθούμε με τον βασικό κανονισμό. Το θέμα ήταν εάν χρησιμοποιούμε δάνεια και εγγυήσει για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, πώς ακριβώς ορίζουμε τις παρατυπίες. Δεν έχω χρόνο για να σας πω όλες τις λεπτομέρειες γιατί ήταν μακρά η συζήτηση. Τέλος πάντων το συμπέρασμα ήταν πως ε, στην ε, Ουγγρική περίπτωση δεν υπάρχει διπλή χρηματοδότηση ή υπερκάλυψη. Διαυκρινίσαμε αυτές τις ε, περιπτώσεις και ελπίζω θα, μπορέ, θα μας επιτραπεί να συνεχίσουμε με αυτή τη λύση. Θα ήθελα τώρα, εν είδη συμπεράσματος, να προσθέσω κάποια πράγματα. Ήταν ε, θετική η εμπειρία αυτών των μεικτών προϊόντων και συστήνουμε να ενισχυθεί ε, περισσότερο ρόλος αυτών των ε, μέσων. Βάσει του βασικού κανονισμού του CPR είναι δυνατή, δυνατός ο συνδυασμός διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, διαφόρων ταμείων, διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Φαίνεται όμως πως ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται ε, να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τα χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε εξετάσει κάποια πρώτα σχέδια και φαίνεται ότι αυτές οι συστάσεις ε, τελικά είναι πιο περιοριστικές και από τον βασικό κανονισμό. Η διαφορά ανάμεσα στην περίοδο 2007-2013 και της επομένης θα είναι ότι είχαμε περιορισμένου κανόνε και σχεδόν καθόλου κατευθυντήρε γραμμέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προηγούμενη περίοδο και αυτό αφήνε μεγαλύτερο περιθώριο λιγμών για τα κράτη-μέλη. Στη νέα περίοδο, αντίθετα, θα έχουμε πιο εξελιγμένο κανονισμό με περισσότερε κατευθυντήριε γραμμέ που δυστυχώς δεν ε, συνάδουν με τις τρέχουσες πρακτικές ε, πάντοτε των κρατών μελών. Όμως ε, το βασικό είναι ο χρονισμός Χρειαζόμαστε εγκαίρως ε, τις ε, απαιτούμενες πληροφορίες ε, και τα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε. Σας ευχαριστώ και θα προσπαθήσω να απαντήσω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Πολύ σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Πολύ ενδιαφέρουσες, εξαιρετικές παρουσιάσεις. Βλέπουμε διαφορετικές απόψεις, όμως η βάση της συζήτησης είναι πάρα πολύ καλή. Συνάδελφοι, ήρθε η σειρά μας. Ερωτήσεις, συστάσεις, παρατηρήσεις. Λουαρ, Κύριε Ρούερ, έχετε τον λόγο, Ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι κατά των χρηματοδοτικών μέσων. Πιστεύουν έχουν κάποια αξία, αλλά βλέπω και ε, κάποια προβλήματα δημιουργούν ε, σε υποδομές ορισμένα μέρη όπου δεν πληρούν και τις... δεν έχουν, φέρει και το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ε, λαμβάνουμε την καλύτερη αξία για τα χρήματα που επενδύουμε βάσει των όσων ε, να επιτύχει η Επιτροπή, πιστεύω. Αυτό που θέλω να πω δεν ε, αντιτίθεται στην περιφερειακή πολιτική. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το σκεπτικό στο οποίο βασίζονται τα χρηματοδοτικά μέσα. Περισσότερο από ότι οι λεπτομέρειε του κανονισμού και συγκεκριμένοι χρηματοδοτικοί κανόνες ή νομικέ δομέ. που δεν μπορώ φυσικά να καταλάβω εγώ ως πολιτικός, έχω μια πιο γενική γνώση του θέματος. Λοιπόν, ε, συνολικά, Αναφέρθηκε η αποτυχία της αγοράς market failure και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η έκφραση, αλλά καταλαβαίνω ότι προσπαθούσατε να πείτε. Ενώσατε κάποια διένεξη μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων Βρετανών και ε, κάποιου βουλευτή ίσως Βρετανού. Καταλαβαίνουμε τι πάτε να πείτε. Αφού που με ανησυχεί είναι η ο κίνδυνος μετατόπισης αυτών των χρηματοδοτικών μέσων, δηλαδή επενδύσεις ε, σε σημεία που δεν χρειάζεται, που δεν το αξίζουν και αφαίρεση χρημάτων από άλλες επενδύσεις. Ε, υπάρχει λοιπόν ένας κίνδυνος ε, ο οποίος κάνει ακόμα πιο δυσδιάκριτη τη διάκριση μεταξύ της δημόσιας επένδυσης που δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης σε αντίθεση με οργανισμούς που επιλέγουν ε, τις πιο επιτυχημένες επενδύσεις. Για το ένα με υπέρ, για το άλλο όχι. Αυτό λοιπόν υπογραμμίζει κατά την άποψή μου την ανάγκη η Κομισιόν να εστιαστεί σε τομεί που χρειάζονται καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα. Ανάπτυξη. Και αναφέρατε και την μικροχρηματοδότηση στην Ουγγαρία. Και αυτό εντάσσεται στην ίδια κατηγορία. Είναι μια χρήσιμη έννοια το να αναπτύξουμε μια αγορά που δεν έχει αναπτυχθεί πλήρω όσον αφορά την καινοτόμο χρηματοδότηση. Αλλά επαναλαμβάνω αυτό είναι κίνδυνο μια επένδυση η οποία φέρνει κάποιο κεφάλαιο το οποίο καταλήγει τελικά σε, μια, ε, σε ένα έργο το οποίο δεν το χρειαζόταν αυτά τα χρήματα τόσο πολύ, το οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αλλού. Περισσότερο παρατηρήσεις κάνω παρά ερώτηση. Πρόεδρος, ε, ναι, ουσιαστικά ξεκινώ τη συζήτηση. Ανοίγω τη συζήτηση, δεν ζητά μόνο ερωτήσεις, αλλά να σας υπενθυμίσω το χρονικό περιορισμό που έχουμε και παρατηρώ και παρακαλώ περιοριστείτε στα δύο λεπτά, αν μπορείτε. Κυρία Μαλέτιτς, ευχαριστώ πολύ. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες σε όλα τα κράτη-μέλη. είναι σημαντικό για τη βελτίωση της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής ε, στο κομμάτι αυτό τη κοινωνίας. Θα πρέπει κάπως να επιταχύνουμε, απλουστεύοντας τις διαδικασίες ε, στα κράτη-μέλη. Με ενδιαφέρει αυτή η περίπτωση της Ουγγαρίας. Ε, αρχίζεται συνδυάζοντας ε, μικροπιστώσεις με δικαιούχους γιατί και στην Κροατία έχουμε περιπτώσεις όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας λαμβάνουν κομμάτια του ERDF για παράδειγμα αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να συγχρηματοδοτήσουν το υπόλοιπο. Λαμβάνουν το 45% για παράδειγμα, αλλά τους λείπει το 65%. Ε, και μερικές φορές τα έργα, ε, ε, κάποια άλλα έργα πλέον δεν είναι επιλέξιμα και πρέπει να τα καλύψουν εξ ολοκλήρου με δικούς τους πόρους οπότε δεν έχουν πρόσβαση στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να λάβουν υποστήριξη από τράπεζε για τα υπόλοιπα αυτά κομμάτια πρέπει να χρηματοδοτήσουν. Οπότε λόγω αυτών των συνθηκών ε, υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης. Θα με ενδιαφέρε να μάθω πώς καταφέρατε ε, να συνδυάσετε, να βάλετε στο παιχνίδι και τη μικροπίστωση, ειδικότερα αφού υπάρχουν οι κανόνες ε, κρατικής ενίσχυσης, έχετε κάποιες συγκεκριμένες ε, συνθήκες, κάποιες προϋποθέσεις για τη μικροπίστη που σας προστατεύουν σε σχέση με αυτούς τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητός, ο κύριος Αουλμπρέχτ. Ναι, δύο παρατηρήσεις και δύο ερωτήσεις. Η μία παρατήρηση είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που ακούσαμε. Αποδεικνύει τι εννοούμε με την έννοια απλούστευση. Έχω με την εντύπωση ότι με τις πρόσφατες αλλαγές η κατάσταση περιπλάκη έχει γίνει πιο περίπλοκη από ό,τι παλιότερα. Έτσι φαίνεται να γίνεται στην Ουγγαρία. Λέμε απλούστευση, αλλά δεν ξέρουμε αν έγινε πραγματικά είναι απλούστεροι κανόνες αλλά είναι πιο περιοριστικοί. Ε, ενδιαφέρουσα αυτή η έννοια υπό την οποία απλούστευση μεταφράζεται σε περιορισμό. Μετά αναφέρατε το πολιτικό νόημα, το τι σήμαιναν πολιτικά οι χρηματοδοτικές ε, ενισχύσεις στην προηγούμενη ε, δημοσιονομική περίοδο. Έβαζαν τα λεφτά σε ένα ασφαλές μέρος ουσιαστικά ε, το οποίο καταγραφόταν ως ταμείο. Θυμάμαι και τη συζήτηση και εδώ στο Κοινοβούλιο ήταν μια από τις ε, λύσεις σε περίπτωση ασάφες. Για να μην χαθούν τα χρήματα τα βάζαμε μέσα σε ένα χρηματοδοτικό μέσο για να είναι ασφαλή. Οπότε το ερώτημα είναι ισχύει ακόμα αυτό. Είναι καλή λύση το να παρκάρουμε έτσι τα χρήματα περιμένοντας καλύτερες εποχές ή Τώρα τα χρησιμοποιούμε ίσως μία φορά. Υπήρχε και αυτός ο κανόνας, ειδικότερα στο πλαίσιο του Τζέσικα. Λοιπόν, αν συμβαίνει αυτό, αν υπάρχει διπλή επιλεξιμότητα, πρέπει να υπάρχει κάποια υποχρέωση τι χρηματοδοτείται μόνο με ενίσχυση και τι με χρηματοδοτικό μέσο. Γιατί είναι σαφές για όλους ότι οι ενισχύσεις είναι πιο ελκυστικές προς τους δικαιούχους γιατί είναι ευκολότερες. Οπότε για τις οικονομίες γενικότερα τα χρηματοδοτικά μέσα είναι καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Για τους τελικούς δικαιούχους όμως αυτοί προτιμούν τις ενισχύσεις γιατί είναι απλούστερες από τα χρηματοδοτικά μέσα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφής διαχωρισμός μεταξύ ενισχύσεων και χρηματοδοτικών μέσων. Και τελευταίο, δεν νομίζετε ότι το ΕΦΣΙ άλλαξε την κατάσταση το Ταμείο Γιούνκερ. Αυτό δεν πιστεύετε ότι άλλαξε την κατάσταση όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βανίσταλρο, δύο λεπτά. Δύο ερωτήσει. Η μία αφορά αυτό το εγχειρίδιο του 2013, 11-12, ανταποκρίνεται στα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει κάποια μελέτη που να αφορά την ε, μετέπειτα περίοδο. Θα ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα να δω αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ του πριν και του μετά. Άλλη ερώτηση. όσον αφορά τις εγγυήσει για τα δάνεια. Εδώ μας ε, λέτε ότι υπάρχουν ε, συνδυασμένες εγγύησει. Και αναρωτιέμαι, είναι θεωρητικό το πρόβλημα. Τα δάνεια αυτά προέρχονται χρηματοδότηση από την Ευρώπη μόνο ή από κρατικές πηγές, ε, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις κοινότητες, τους δήμους. Μπορεί να προκύψουν προβλήματα ή όχι. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ελπίζω να μην υπάρχουν βασικά προβλήματα, αλλά ίσως να υπάρχουν. Η κυρία Βάνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους τρεις εμπειρογνώμονες για τις εξαιρετικές τους παρουσιάσεις. Οι πράσινοι θέλουν να στηρίξουν και νοτομίες και ενδεχομένως ε, και στο παρελθόν είχαμε εκφράσει τις ε, αμφιβολίες μας όσον αφορά τη δυνατότητα χρηματοδότησης τέτοιων καινοτόμων πρωτοβουλειών μέσω των ε, χρηματοδοτικών αυτών μέσων. Η ερώτησή μου αφορά ένα πάρα πάρα πολύ, αν θέλετε, σημαντικό τομέα. Διαφάνεια και δημοκρατικός έλεγχος. Αν όντως υπάρχει μία τακτική και εντελεχής διαδικασία ελέγχου Πώς διασφαλίζετε ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι ακριβή. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό ε, είναι και το θέμα του ποσοστού απορρόφησης ε, εκταμίευσης ε, μέσω αυτών των μέσων και ξέρουμε ότι το, λογιστικό, το ελεγκτικό συνέδριο έχει πάρα πολύ αρνητική αξιολόγηση. Πώς μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά τις πληρωμές. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στη γνωμοδότηση αυτού ελεγκτικού συνεδρίου 2012 για την περιφερειακή πολιτική και πριν από λίγους μήνες βλέπουμε ότι αυτή η χρήση των ε, χρηματοδοτικών αυτών μέσων για την ε, γεωργική πολιτική και αυτό που πολύ φοβάται ή ανησυχεί τον κύριο Όλμπρεχτ, πολύ φοβάμαι ότι φαίνεται από την μελέτη που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο. Βλέπουμε ότι η χρηματοδότηση τελικά περνάει μέσα από αυτές τις δυνατότητες και ουσιαστικά βοηθάει αυτούς οι οποίοι τελικά εποφελούνται και αυτοί που θα έπρεπε να είναι οι δικαιούχοι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραδείγματος χάριν, δεν φτάνουν μέχρι αυτούς τα κονδύλια αυτά τα οποία παραμένουν στις τράπεζες και δεν χρησιμοποιούνται από αυτούς που ε, ουσιαστικά και δικαιολογημένα θα έπρεπε να μπορούν να υποφεληθούν. Είδαμε λοιπόν ότι το κύριο πρόβλημα είναι η περιπλοκότητα των διαδικασιών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι αυτήν την πηγή χρηματοδότησης και επαναλαμβάνω οι πιστώσεις αυτά, τα κονδύλια αυτά παραμένουν στις τράπεζες. Ουσιαστικά βοηθούν στην ε, καλύτερη οικονομική κατάσταση των τραπεζών, έτσι ώστε τα κεφάλαιά τους να είναι αρκετά. Και σήμερα βλέπουμε ο τραπεζικός τομέας θα πρέπει πραγματικά να βοηθήσει την πραγματική οικονομία, να τροφοδοτήσει αυτούς που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα γνωρίζει σήμερα το πρόβλημα και σίγουρα υπάρχουν σήμερα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Γερμανία που οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με χαμηλότερα επιτόκια και με ε, πιο απλές διαδικασίες. Το θέμα είναι αυτές οι τόσο περίπλοκες διαδικασίες να πάψουν να αποτελούν εμπόδιο γιατί αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα τελικά δεν χρηματοδοτούν εκεί που ε, θα έπρεπε αρχικά, δεν στοχεύουν τους τομείς αυτούς της οικονομίας για τους οποίους σχεδιάστηκαν. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε όλους αυτούς που έχουν και τα τυπικά προσόντα αλλά και ανάγκη από αυτή τη χρηματοδότηση να έχουν πρόσβαση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα της απορρόφησης αυτών των κονδυλίων. Οι εκταμιεύσεις που γίνονται, οι πληρωμές που γίνονται είναι πολύ κάτω από τα ποσοστά που θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας, ε, ώστε να απαντήσουν, να σχολιάσουν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες. Όσον αφορά τα ωφέλη, ίσως να ήμουν ε, λίγο υπερβολικά συνοπτική στην παρουσίασή μου στην προηγούμενη αλλά και στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο προσπαθούμε να εμπλέξουμε περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα να αποδεσμεύσουμε το δυναμικό που υπάρχει εκεί στην οικονομία. Αυτό είναι ένα από τα ωφέλη που φέρνουν αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα, αλλά είναι η μόχλευση Δηλαδή για κάθε ένα ευρώ του ESIF μέσω των χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να υπάρξει και περισσότερη δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση. Κάτι άλλο που αφορά ορισμένα κράτη-μέλη. Τίθενται τα ερωτήματα την επόμενη φορά θα πάρουμε τόσα, θα πάρουμε καθόλου. Τα χρήματα αυτά επανέρχονται για επαναχρησιμοποίηση ουσιαστικά επιβάλλουν μεγαλύτερη πειθαρχία σε όλους τους συμμετέχοντες και αυτό με φέρνει στο άλλο ζήτημα που τέθηκε από πολλούς εδώ αυτό που δεν θέλαμε να συμβεί πουθενά αυτή τη φορά ήταν ήταν ε, τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα να μην χρησιμοποιηθούν επαρκώς. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αξιολόγηση στην αρχή της ε, προγραμματικής περίοδου Κάποιες διαχειριστικές αρχές παραπονέθηκαν λέγοντας «Α, ακόμα διοικητικός φόρτος είναι πολύ περίπλοκο, θα πάρει πολύ χρόνο». Αλλά τώρα μας λένε τελικά ότι μας βοήθησε να δούμε τις αγορές, να δούμε τι συμμετοχή υπάρχει, τι δυνατότητα συμμετοχής υπάρχει από τον ιδιωτικό τομέα, κατά πόσο χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το θέμα των επιτοκίων. Επίσης, μας ανάγκασε να δούμε κατά πόσο χρειάζεται συνδυασμός ε, με τις ενισχύσεις και να επιβεβαιώσω είναι δυνατόν και οι σκέψει αυτές ε, να μην υπάρχει διπλή χρηματοδότηση είναι πολύ σημαντικέ. Αυτό το λέει και ο οικονομισμός. Και εμείς από πλευράς Κομισιών ανησυχούμε για το κατά πόσο συνδυασμό τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στο να αιτείται κανεί ε, ε, βάσει άλλων κανόνων για άλλο μέσο. Υπάρχει δυνατότητα περιπλοκής, επιπλοκής της κατάστασης. Αλλά και σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν παραδείγματα όπου με ξεχωριστούς μηχανισμούς λογιστικούς μπορεί κανείς να αντλήσει χρήματα και από τα δύο. Για το ΕΦΣΙ τώρα είναι ένα νέο στοιχείο από την εθέτηση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Εμείς προσπαθούμε να φροντίσουμε να είναι συμπληρωματικό με το ΕΦΣΙ ε, ε, ε, και με το Horizon. Το SF όπως χρησιμοποιείται συμπληρώνει και ένα μεγιστοποιητή μόχλευση, αντιμετωπίζει τα προβλήματα Όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, να εξηγήσω λίγο τίθε το θέμα της διαφάνειας και του δημοκρατικού ελέγχου. Αυτό είχε αλλάξει την σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, δεν υπήρχε τόση διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο δημοσιεύεται μέχρι την 1η Οκτωβρίου μια ετήσια σύνοψη που συγκεντρώνει πληροφορίες για κάθε χρηματοδοτικό μέσο που υποστηρίζεται στο πλαίσιο του ERDF και του ESF. Από του χρόνου ε, θα το λάβετε το πρώτο για την νέα περίοδο 1η Νοεμβρίου. Οπότε θα έχετε δύο από του χρόνου. Η μεθοδολογία πληρωμής, ε, το είπατε πολύ σωστά, είναι ένα βασικό σημείο προβληματικό για την προηγούμενη περίοδο. Οι αρχές έβαλαν 100% τα χρήματα μέσα και μετά αυτά κάτσαμε στο ταμείο και αυτό αποτέλεσε αντικείμενο επικρίσεων και ε, τέθηκαν ερωτήματα για το κόστος σύμφωνα με τον νέο κανόνα, ε, μια πρώτη πληρωμή στο ταμείο πρέπει να δηλωθεί ε, στην Επιτροπή, αλλά η διαχειριστική αρχή δεν μπορεί να δηλώσει περισσότερα έω ότου τα ταμεία αυτά, τα κονδύλια αυτά έχουν φτάσει στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Υπάρχουν κάποια ποσοστά δηλαδή. Έχουμε ένα ε, σημείωμα με κατευθυντήρια γραμμέ αν θέλετε να μάθετε περισσότερα. Υπάρχουν ποσοστά. Σκοπός είναι να φτάνουν τα χρήματα στην αγορά. Το συζητήσαμε με τα κρατημένη και το Κοινοβούλιο. Ο σκοπός είναι να φτάσουν τα χρήματα στον δικαιούχο. Και μετά ε, και όλο το ζήτημα των κατευθυντήριων γραμμών της απλούστευση τέθηκε από τους συναδέλφους και τους ε, και βρεθήκαμε και εμείς και η Κομισιόν σε μια περίεργη κατάσταση διότι ξεκινήσαμε όλη αυτή την περίοδο λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ε, ολοκληρωμένους κανόνες, ένα σαφές πλαίσιο το οποίο έχει υιοθετηθεί από τους ε, συνομοθέτες και εσείς κρατημέλη είστε ένας από αυτούς και δεν θέλουμε άλλες κατευθυντήριες γραμμές γιατί θεωρούμε ότι είναι σαφές τώρα. Αυτό ε, ήταν ο σκοπός μας, αλλά όπως το παρατηρήσετε αυτό δεν κράτησε πολύ, γιατί ε, αμέσως μας ε, έστειλαν ένα σωρό ερωτήσεις, σχόλια και το θέμα αυτό του οικονομικού ελέγχου στην προηγούμενη περίοδο αποτέλεσε ένα πρόβλημα. Πολύ δύσκολη ήταν η έλεγχη, διάφορα ζητήματα τα οποία σαν πολλά προβλήματα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε για να απλουστεύσουμε τα πράγματα ήταν να, να δώσουμε διευκρινιστικές κατευθυντήρες γραμμές. Αυτό που λέγαμε δεν είναι ήπια Αυτή τη φορά δεν έχουμε ήπια νομοθεσία. Υπάρχει νομοθεσία. Έχει θεσπιστεί. Έχουμε και μια επιτροπή εμπειρογνωμών των κρατών μελών, όπου τα κράτη-μέλη επανέρχονται εκεί και γίνονται κάποιες ζωηρές συζητήσεις και καταλήγουμε σε μια έκδοση που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας και παρέχει συμβουλές, διευκρινήσεις, αλλά ταυτόχρονα αν οι διαχειριστικές αρχές, αν τα κράτη-μέλη θέλουν να φτιάξουν ένα δικό τους οργανισμό, σύμφωνα με την νομοθεσία, αυτό τελικά είναι το σημαντικότερο. Ακούσαμε όλα για την απλούστευση. Έχουμε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου όπου θα συζητά για τα χρηματοδοτικά μέσα και για να κλείσω από πλευράς μας το σημαντικότερο είναι τελικά να είναι απλό για τον τελικό δικαιούχο, ακόμη και αν σε υψηλό επίπεδο είναι περίπλοκο, γιατί τα δημόσια κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε τελική ανάλυση, η μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει να μπορεί να έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζεται. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα, αλλά ήταν πολλά τα ζητήματα που έπρεπε να απαντήσω και ενδιαφέροντα. Uh, Ευχαριστούμε, κύριε Ράους. Ε, ε, ε, θα είμαι σύντομος. Πρώτον, για τον οικονομικό έλεγχο, όντως υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο οικονομικών ελέγχων, δηλαδή υπάρχει μεγάλο άγχος από πλευράς των κρατών σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων ε, και δύσκολα βλέπουν τις συμβουλές ως μόνο γραμμές, διότι για τον οικονομικό έλεγχο στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραδείγματο χάρη, ε, μιλάνε για κατευθυντήριες γραμμές και προσπαθούν να τα φορτώσουν όλα σε αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Είναι χρήσιμα αυτά που ακούσαμε. Πιστεύω πάντως πως το μόνο που θα μπορούσε να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα στο μέλλον είναι να απαντάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ε, τίθενται τέτοια ζητήματα. Θα μας βοηθούσε πολύ αυτό στο μέλλον. Δεύτερον, σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για το, το κλειδί είναι οι εμπορικές ε, αποφάσεις, δηλαδή οι αποφάσεις των εμπορικών τραπεζών κυρίως ε, για τα νέα χρηματοδοτικά μέσα και το θέμα των αμοιβών ε, φυσικά έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος. Αυτά. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Νίκολς, θέλετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για τις ερωτήσεις. Θα ήθελα ε, να μου επιτρέψετε να σας πω ακριβώς τι γίνεται στην πράξη. Για την, λήψη αποφάσεων πρέπει να υπολογιστεί το ποσό του δανείου και σας είπα το 10% ήδη η δηλαδή ε, συνυπολογίζεται εξ ορισμού και μετά το, το υπόλοιπο κενό, αν θέλετε, το υπολοιπόμενο ποσό θα καλυφθεί βάσει των ε, κανονισμών. 10% λοιπόν ήδη οι και μετά το πρόγραμμα. Αν είναι βιώσιμο το πρόγραμμα που προτείνεται, παίρνουμε ε, αυτή την μικροπίστη και αν υπάρχει και επιδότηση συνυπολογίζεται, συνδυάζεται. Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες βάσει και των δύο ε, αυτών μηχανισμών ποτέ δεν ξεπερνούν φυσικά το 100% της επένδυσης. Συζητήσαμε εκτενώς το θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα των οικονομικών ελέγχων και συμφωνήσαμε και εντοπίσαμε το πρόβλημα. Το διευκρινίσαμε όμως και προκύπτει, όπως σας έλεγα προηγουμένως, ότι μπορούμε να ε, συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το σύστημα. Για τις κρατικές ε, προμήθειες, το de minimis χρησιμοποιούμε και... Φροντίζουμε να μην παραβιάζουμε τις, ε, τους όρους για τις κρατικές προμήθειες, τις εξαιρέσεις δηλαδή. για το, ε, τη, τη μη χρήση των κονδυλίων Δεν είναι δυνατόν ε, στα πλαίσια αυτού του συστήματος να παραμένουν τα χρήματα ή στην τράπεζα ή σε κάποιο άλλο ε, στάδιο και να μην δίνονται στις επιχειρήσεις. Μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτό το νέο σύστημα, αυτό είναι θετικό. Όμως ε, θεσμικά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, γιατί παλιότερα χρησιμοποιούσαμε το θέμα της αναχρηματοδότησης. Ε, επαναχρησιμοποίηση των επενδύσεων και με την ε, μεταρρύθμιση δεν ξέρω τι θα είναι δυνατόν. Επίσης, μεθοδολογία για το κόστος και τι αμοιβέ ε, πάντα δείχνει το ζήτημα των κανονισμών των κρατικών προμηθειών. Οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την επόμενη περίοδο με το ίδιο σύστημα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you very much for the excellent... Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τι εξαιρετικέ παρουσιάσεις, τις απαντήσεις σας, τη συζήτηση. Εγκρίναμε και τις αποφάσεις σήμερα το πρωί των συντονιστών. Στα διάφορα υπάρχει κάτι, ναι. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Μάλατιτς να πει κάτι για τις προφορικές ερωτήσεις. Η κυρία Μάλατιτς για τις προφορικές ερωτήσεις όσον αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών της ε, πολιτικής συνοχής. Είμαι στο τέλος του 2015 και καταρχήν οι δεσμεύσεις για το έτος 17 ή 18 εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα προοδεύσει η διαδικασία στην κάθε χώρα, για την κάθε χώρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε με την Επιτροπή ποιος μηχανισμός μπορεί να υλοποιηθεί εδώ έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ε, εφαρμογή και να αποφύγουμε την αποδέσμευση. Πιστεύω ότι η Επιτροπή ήδη έχει κάποιες ε, αντιρρήσεις όσον αφορά τις δεσμεύσεις που θα λάβουν χώρα τέλος του 2015 είναι όμως σημαντικό να δούμε τι δεν λειτουργήσε, ποια ήταν τα βασικότερα εμπόδια για αυτήν την ε, περίοδο και να αποφύγουμε κάτι παρόμοιο στο τέλος του 17 και στο τέλος του 18. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ναι, θα το συζητήσουμε εξ ονόματος της Περιφερειακής Επιτροπής. Αυτό μου λέτε τώρα, έτσι αυτή την προφορική ερώτηση. Εντάξει. Οκ, θα ακολουθηθεί η κανονική διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνεδρίασή μας τον Ιανουάριο. Σας εύχομαι καλή και επιτυχημένη περίοδο μέχρι τις διακοπές. Τις ευχές μας και στους διερμηνείς σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος της συνεδρίας.